Okay, dear colleagues, please do sit down. We will start. Καθίστε συνάδελφοι. As our chair, Mr. Lavia. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Λαβία, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις σήμερα. Θα τον αντικαταστήσω. Αν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο. Σήμερα το πρωί. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Uh, Οι πράσινοι ζήτησαν την προσθήκη ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτινόμενης κατεξοδότηση πράξης για εξαίρεση του καδμίου. Ε, κανονικά το είχαμε τελευταίο σημείο αύριο το πρωί. Αν έχετε αντιρρήσεις όσον αφορά το αίτημα των πρασίνων, πείτε το μου. Η δεμή θεωρώ συγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Άλλο σημείο. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ακρόαση για το να σταματήσουν οι, ζωντανοί οι τομές στα ζώα. Η Ήτρε, η Έμβη και η Πέτη μαζί, θα συνεδριάσουμε μαζί τους τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα ΖΑΝ 4Q2, εδώ δηλαδή. Και όλα τα μέλη καλούνται να παραστούν, είναι σημαντικό θέμα, είναι η πρώτη πρωτοβουλία πολιτών που θα συζητηθεί στην Επιτροπή. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να συμμετάσχετε στην ακρόση για να, σταματήσει, να σταματήσουν αυτά τα πειράματα και το μέσα στα ζώντα ζώα. στην ε, μήνυ ολομέλεια του Μαΐου θα γίνει συνεδρίαση έκτατη στη συνεδρίαση του στη Σύνοδο στις 18 Μαΐου στο Στασβούργο στις 7 το απόγευμα θα γίνει έκτακτη σύνοδος μας 7 το απόγευμα 18 Μαΐου Δευτέρα ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σεύκοβιτ συζήτηση όσον αφορά τον διαθρωμένο διάλογο. Θα συζητήσουμε διάφορα θέματα. Οπότε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας σας συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ε, υπάρχει αλλαγή στη γραμματεία της Επιτροπής ΕΝΒΗ, Μασότο Ρονού. Ε, έρχεται από την Επιτροπή Γεωργίας και συμμετέχει από 1η Μαΐου στη γραμματεία μας. Την καλωσορίζω λοιπόν. και την ευχαριστώ για τη βοήθεια που θα μας δώσει. Διερμηνία. Έχουμε 21 γλώσσες. Όσοι συνήθως. Εξεργούνται τα μαλτέζικα, τα ογοδελικά και τα αστωνικά. Και οι εξεκτονικές συνεδριάσεις θα υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελο μέσω του e-meeting. Και η συνεδρίαση εκπέμπεται στο διαδίκτυο για τους ενδιαφερόμενους για τα θέματα μας. Τρίτο σημείο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 23ης και 24ης Φεβρουαρίου Υπάρχουν μήπως αντιρρήσεις. Αν έχετε αντιρρήσεις, παρακαλώ γνωστοποιήστε τες στην γραμματεία μέχρι το τέλος συνεδριάσεως. Αν δεν προβληθούν ενστάσεις μέχρι το τέλος συνεδριάσεως, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Σημείο 4. Έχουμε το σχέδιο εκθέσεως που αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα. Σημαντικό θέμα. Καταρχάς να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Φρανσουάς Γκρόστετ. Έχετε το λόγο όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχουμε να συζητήσουμε σήμερα το πρωί πράγματι την αναθεώρηση του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα, μια έκθεση ιδιαίτερα εκτεταμένη και έχω κάποια σημεία να θίξω που τα θεωρώ σημαντικότατα. Θέλω να τονίσω τρεις προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της αντιστάσεως στα αντιβιωτικά, μεγάλο διακύβευμα για τη δημόσια υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιες προτάσεις σχετικά με αυτό, αλλά θεώρησα ότι δεν είχε προχωρήσει αρκετά. Προτείνω να απαγορευτεί η χρήση σε προληπτικά των αντιβιωτικών, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν γίνεται μια χειρουργική επέμβαση, φερρυπίν, και πρότεινα και το 107 να διευκρινιστεί το άθρο όσον αφορά τη συνταγογράφηση και την πώληση, να ενθαρρυνθεί η έρευνα επίσης στο τομέα της θεραπείας με αντιβιωτικά και να εισαχθεί και η έννοια της αμοιβαιότητας, ούτως ώστε οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα αντιβιωτικά στην Ευρώπη να εφαρμόζονται και στα τρόφιμα και το κρέας που εισάγεται για κατανάλωση. Είναι ένα θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και μπαίνοντα τώρα σε λεπτομέρειε, θεωρώ ότι απαγορεύεται η πώληση αντιβιωτικών στο διαδίκτυο online και κυρίω των κτηνιατρικών ε, φαρμάκων. Στεγγράφηση. Η πώληση στο διαδίκτυο διευκολύνει τι απάτε, την παραποίηση των προϊόντων, περιπλέκει την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων. Αυτή η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων είναι κάτι που είναι κρισίμου σημασία όσον αφορά την παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιωτικών παρά τους φραγμούς που προτάθηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση των κινδύνων αυτών, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αποτελεσματικούς ελέγχους και γι' αυτό πρότεινα μια συνολική απαγόρευση, γενική απαγόρευση. Στην πρώτη συζήτηση που διεξήχθη, η μεγάλη πλειοψηφία από εσά συμφωνούσατε με αυτή την αρχή, ακόμα και αν γνωρίζω ότι ακολουθούνται σε κάποια, κάποια, κάποια μέλη, ε, κάτι μέλη κάποιες πρακτικές που διευκολύνουν την πόλη. Πρέπει να είμαστε λογικοί να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να περάσουμε μέσω απαγορεύσεως. Δεύτερο σημείο, πρέπει να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την καινοτομία πραγματετομέας των κτηνιατρικών φαρμάκων αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα διαθεσιμότητας προϊόντων σε κάποιες αγορές και για κάποια είδη. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα και δυσκολία. Η έρευνα έχει μείνει πολύ πίσω διότι δεν υπάρχουν, δεν είναι πολύ ελκυστικό ο τομέας για τα διάφορα εργαστηρία και έχουμε πρόβλημα εκεί διαθεσιμότητας φαρμάκων. Εξ αυτού λοιπόν πρότεινα να επεκτείνουμε την περίοδο, να παρατείνουμε την περίοδο προστασία των νέων αντιβιωτικών στα 18 χρόνια αντί τα 14 χρόνια και να παρατείνουμε σε ένα από συν ένα σε σύν δύο χρόνια την αρχική προστασία σε περίπτωση της προστίκης ενός σημαντικού είδους. Ε, αν θέλουμε λοιπόν να γίνει κάτι καινούριο σε αυτή την καινοτομία θα πρέπει να δώσουμε αυτή την όθηση που είναι σημαντική. Η δεμή θα εξακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες δυσκολίες προτείνω περίοδο προστασίας 5 ετή, μη σωρευτική, για κάποιες νέες μελέτες ή νέες δοκιμές, μετά την αδειοδότηση, για τη διευκόλυνση ανάπτυξης ή βελτιώσεως υφισταμένων προϊόντων, ε, για πρόδρομο σωσής ή γενώσιμα φάρμακα. Η δημόσια υγεία και θεσιμότητα των προϊόντων, ας μην ξεγελιόμαστε, είναι αλληλένδετα, άρρηκτα συνδεδεμένα. Επιμένω επ' αυτού θα επιμείνετε επί του κόστου των προϊόντων, το κατανοώ αυτό, αλλά η αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων δεν είναι η αγορά των άλλων των φαρμάκων προς ανθρώπινη κατανάλωση, δεν υπάρχει η ίδια μορφή της αγοράς, πρέπει να υπόψη και η βιομηχανία των γενοσύμων ε, έχει κάθε συμφέρον να υπάρχει καινοτομία, υπάρχει καινοτομία, θα υπάρχουν και περισσότερα γενώσιμα φάρμακα μετά. Η βιομηχανία χρειάζεται προβλεψιμότητα. Σκεπτόμενοι όλα αυτά, υποβάλλω τις σχετικές προτάσεις. Τρίτη προτεραιότητα, η βελτίωση της ε, φαρμακοεποπτείας, της εποπτείας των φαρμάκων, ξεκίνησε από την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδραζόταν επί της επισημάσεως και του εντοπισμού των ε, κινδύνου. Είναι μια πρόταση που την υποστηρίζω, θα μειωθεί η γραφειοκρατία με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται μια νέα ισορροπία. Θα πρέπει τακτικά να υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις όσον αφορά τον έλεγχο των φαρμάκων τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της ζωής του προϊόντος όταν οι συνέπειες της χρήσης σε μεγάλη κλίμακα ε, δεν είναι πολύ γνωστές. Από τη στιγμή που ένα προϊόν είναι γνωστό, όταν θα έχουμε μπορέσει να το κρίνουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό κλπ, ή ποιους κινδύνους δημιουργεί, εκεί θα μπορέσουμε να προβλέψουμε ε, να έχουμε εκθέσει προβάλλονται σε λιγότερα τακτά διαστήματα. Λοιπόν πρέπει τα πρώτα χρόνια να προσέχουμε τι γίνεται με κάποιο φάρμακο και εν συνεχεία το σύστημα μπορεί να χαλαρώνει στον αφορά την παρακολούθηση. Θέλω να επανεισαχθεί η έννοια της λήξης της αδειοδότησης στην αγορά, ακύρωσης μάλλον, για να βοηθηθεί μια πολύ καθυστερημένη διάθεση στην αγορά χωρίς επικαιροποίηση λόγω νέων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για ένα φάρμακο υπάρχουν κάποια φάρμακα που δίδονται, κάποιες άδειες που δίνονται κάποιο φάρμακο που δεν έχει ε, διατεθεί στο εμπόριο και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ισχύει επαόριστον μια αδιαδότηση. Εάν το προϊόν δεν έχει διατεθεί στο εμπόριο σημαίνει ότι τελικά δεν είναι απαραίτητο. Οπότε, τη αυτή περιπτώση θα πρέπει να επανεισαχθεί η έννοια της λήξης ισχύω ε, μιας ε, ε, αδειοδότησης. Αυτές είναι τις προτεραιότητες Υπάρχουν και άλλοι βασικοί άξονες βέβαια που αναφέρω στο σχέδιο της έκθεσης που θεωρώ εξίσου σημαντικούς και πιστεύω και εσείς συμφωνείτε, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη το θίξαμε την προηγούμενη φορά. θέμα να αποφύγουμε να γίνονται ε, συνεχείς διαδοχικές επαναξιολογήσεις που θα παρεκκλίνουν όσον αφορά τον επικίνδυνο χαρακτήρα, τον, ε, την επικινδυνότητα των ουσιών. Ζητώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δύο χρόνια να μας κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τη δυνατότητα να, υπάρχει, να γίνει ε, υποχρεωτικό ένα σύστημα αξιολογήσεως περιβαλλοντικής, δηλαδή αξιολόγηση ε, μοναδικής των ε, ουσιών και όχι κάθε προϊόντος. Στην πρώτη συζήτηση το ανέφερα αυτό και είχα την εντύπωση ότι τότε η πλειοψηφία ήταν υπέρ του συστήματος αυτού. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό αφορά την εναρμόνιση των συνοπτικών παρουσιάσεων των ε, χαρακτηριστικών των προϊόντων. Ε, αν θέλουμε να υπάρξει εναρμόνιση, μεν, μια εναρμόνιση κατά τάξη προϊόντων που θα προσωμείωζε τα προϊόντα μεταξύ τους θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός τότε θα βασιζόταν αποκλειστικά στις τιμές και όχι ε, στις ουσίες και θα ήταν εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να παίξουν πολύ στο περιθώριο κέρδους. Λοιπόν, θέλω ανταυτού να έχουμε εναρμόνιση συνθήκων χρήσεως των προϊόντων που θα ήταν ένα πρώτο βήμα αυτό προς την κατεύθυνση τη σωστή. Τρίτο σημείο που το θεωρώ σημαντικό είναι οι χρήσει εκτός των συγκεκριμένων αδειών. Θα πρέπει να το επαγρυμίσουμε, το προσέξουμε, διότι μια τέτοια χρήση κυρίως των ανθρωπίνων φαρμάκων για τη χρήση στα ζώα ε, έχει διπλό πρόβλημα. Δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και αποθαρρύνονται οι προσπάθειες καινοτομίας. Είναι πολύ εύκολο να λέμε δεν υπάρχουν γενετικά φάρμακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φάρμακο για τους ανθρώπους. Νομίζω δεν είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο διότι δεν δίνουμε κίνητρα για έρευνα και καινοτομία και γι' αυτό ήθελα να έχουμε μια αυστηρή ιεράρχηση των διαφόρων ειδών προϊόντων που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός φαρμάκου. Και η χρήση ενός ανθρώπινου φαρμάκου, φαρμάκου ή τον άνθρωπο θα είναι η τελευταία γραμμή άμυνας. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική καλύτερη. Ε, Έσχατη λύση θα πρέπει να είναι. Τέλος, το θέμα της πωλήσεως ε, της χονδρικής, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει απελευθέρωση των διδοτήσεων της πωλήσεως στη χονδρική. Προτείνω εναρμόνιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των διανομέων του τομέα της χονδρικής και να εναρμονιστούν και κυρώσει σε περίπτωση μη σεβασμού της νομοθεσίας. Γιατί για να αποφύγουμε κίνδυνο αθέμη του ανταγωνισμού αν έχουμε διαφορετικές διατάξεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Εν τη αυτή περιπτώση θα παίζεται κάποιο παιχνίδι από τους χονθρεμπόρους ε, όσον αφορά θα παίζουν μεταξύ των διαφόρων χωρών. Τελευταίο, οι, οι αιτήσει αδειοδοτήσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις. Και εκεί προτείνω απλούστευση της διαδικασίας θα πρέπει να επιτρέπει αντίδραση επαρκή όταν επικρατούν ιδιαίτερες περιστάσεις, αν έχουμε μια επιζωτία φερρυπίν, που θα δικαιολογεί ταχεία διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων. Για να δίνεται άδεια για διάθεση των προϊόντων αυτών σε αυτές τις περιστάσεις, εξαιρετικές περιστάσεις, τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ε, χρήσεως προσωρινής καταρχάς του προϊόντος επιτόπου θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται εν συνεχεία για την υποστήριξη μιας αδειοδοτήσεως μονίμου του φαρμάκου για να αποφύγουμε την επανάληψη δοκιμών που θα μπορούσαν να είναι άχρηστες δοκιμών στα εργαστήρια. Μιλάμε για πλούστευση και πάλι. Να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και να μειώνουμε και το κόστος σε δύο σελίδες ε, συνόψεις, 150 ε, τροπολογίες ε, που συνέταξα. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Δύσκολο να προβάλλω πλήρη σύνθεση. Ήθελα στις εξηγήσεις μου να τονίσω τα ουσιώδη της αναθεωρήσεως, αυτά που θεωρώ εγώ ουσιαστικά και με τα χαράς να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε καταρχάς τις απόψεις των σκιωδών με πρώτο τον εκπρόσωπο του Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας. Ο κύριος Τανασέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και για το έργο της και για την πολύ καλή συνεργασία είναι ευρύτατο το πεδίο του σχεδίου έκθεσης και καλύπτονται μεγάλο μέρος των δικών μου ανησυχιών, έξω και θα περιοριστώ μόνο σε συγκεκριμένα στοιχεία. Στο πλαίσιο της διατήρησης όλων ε, των διάβλων έγκρισης ε, τη κυκλοφορία φάρμακων και για την καλύτερη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, νομίζω ότι οι επιχειρήσει θα έπρεπε να έχουν περισσότερα κίνητρα ε, για να υπαχθούν σε αυτή τη ε, διαδικασία, σε ό,τι αφορά τη διανομή κατά των ιατρικών προϊόντων, υπάρχουν σημαντικές προτάσεις. Και σε ό,τι αφορά την αίτηση, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός της ονομασίας τη δραστική ουσία ή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Είμαι επίσης υπέρ των μέτρων που προτείνονται για τη μείωση της ε, αντοχής ε, στα αντιβιωτικά και σε ό,τι αφορά την πόλη στο Φρόνικο στο ίτερο σχετικά σχετικές προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι κτηνοτροφικές πρακτικές συνεισφέρουν στην περαιτέρω ενίσχυση αυτού του φαινομένου της αντιμικροβιακής αντοχής. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε τη χρήση των φαρμάκων αυτών, των αντιμικροβιακών, ως μια συνήθεια δικασία στα αγροκτήματα. Καλό είναι επίσης να έχουμε πληροφορίες για τα είδη της νόσους που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά και τη μορφή της θεραπείας που ακολουθήθηκε. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει και το πρόβλημα των τρίτων χωρών να λυθεί σε ό,τι αφορά δηλαδή τα αντιμικροβιακά φάρμακα για να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία. Όπως έχω προαναφέρει θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το γεγονός ότι η ε, τροφές που χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές θα μπορούσαν να μπουν στην τροφική αλυσίδα, αν όμως τα κράτη-μέλη έχουν καθορίσει μια περίοδο απόσυρσης. Επίσης, συμφωνώ με τη δυνατότητα εταιρείε να μπορούν να προσθέτουν σχετικές πληροφορίες για λόγους ασφάλειας στη συσκευασία του φαρμάκου. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης των συστημάτων συλλογής των ε, κρατών μελών. Επειδή βέβαια έχουμε επίδραση και στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου και του ζώου, είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την ε, διάθεση των χρησιμοποιητών ε, φαρμάκων ή αυτών που έχουν λήξει. Σε ό,τι αφορά την προστασία των τεχνικών εγγράφων, θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ αφενός καινοτομία, διαθεσιμότητας και αφετέρου προσιτή τιμή κτηνιατρικών φαρμάκων ή προϊόντων. Η συγγύτρια προτείνει να αυξηθεί η αδεία της συγκλωφορίας ισχύς από τρία σε προτεινει να αυξηθει η αδεια τη κυκλοφορία ισχύει από 3 σε 5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να αποβαθμίσουμε τα πρότυπα ασφάλεια. Στηρίζω λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν σχετικά και εμένω στην τριετή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία 42 που προβλέπει περίοδο προστασίας των τεχνικών εγγράφων για τη φτάμενα προϊόντα, εκεί συμφωνώ. Για τη χρήση ενώσιμων δεν θα ήθελα να μπει στο ίδιο επίπεδο η χρήση ανθρώπινων ε, φαρμάκων, μάλλον για τον άνθρωπο, με τη χρήση άλλων εναλλακτικών φαρμάκων που χρησιμοποιηθούν και στα ζώα και γι' αυτό θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες για να αποθαρρυνθεί αυτή η πρακτική. Τα φάρμακα που προσδίδει για τον άνθρωπο ως τελευταία ε, λίστα πρέπει να χωρικούνται. Επίσης για τη μονογραφία, το σύστημα μονογραφίας ε, για τα τενετρικά φάρμακα. Επίσης θέλω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες σχετικά και τέλος το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ, η εναρμόνιση ανά κατηγορία Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρονται και τα παρόμοια ιατρικά φάρμακα ή προϊόντα. Ευχαριστώ των προϊόντων. Ναι, επόμενος ο ο κύριος ε, Πίτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γκροστέτ. Ήταν τεράστιο το έργο που ανέλαβε, πολύπλοκο και το θέμα δεν ήταν και εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ρυθμιστεί ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να ρυθμίσουμε, Δεν ό,τι τι τις ονομασίες. Το θέμα δεν είναι μόνο το ιατρικό φάρμακο ή προϊόν, όπως ε, μπορούμε να διαβάσουμε στην τροπολογία 7. Υπάρχουν και άλλες πτυχές. Ανοσολογία, συνταγογράφηση κτλ. κτλ. Και αυτό μπορεί να αφορά οποιαδήποτε συνταγή για, από οποιονδήποτε κτηνίατρο. Υπάρχουν επίσης κάποιες βασικές έννοιες που δεν ορίζονται παρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Έτσι θα αποφύγουμε σύγχυση σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Βέβαια, πάντοτε σε εύλογα όρια για την εφαρμογή των προϊόντων αυτών, τη χρήση αυτών των προϊόντων. Όλα αυτά ρυθμίζονται στάδια κυκλοφορίας των βασικών παράδειγμα που είναι τα αντιβιωτικά. Χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Και γι' αυτό καλωσορίζω οποιοδήποτε μέτρο ενθαρρύνει τις κεντρικές διαδικασίες, γιατί έτσι διευκολύνεται ένα κοινό σύστημα ελέγχου της πρόσβασης. Υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Δραστικές ουσίες για παράδειγμα. Και τι ρόλο έχουν στα κτηνιατρικά φάρμακα. Ιδίως ότι αυτό το σύστημα μονογραφίας που θεωρώ ενδιαφέρον ως ιδέα. Μια νέα ιδέα που όμως δύσκολα μπορεί να ρυθμιστεί αλλά ευρέως δεδομένη θεωρείται, είναι οι πωλήσει στο διαδίκτυο. Αυτές οι πωλήσει, οι ηλεκτρονικές πωλήσει, ιδίω συνταγογραφούμενων φαρμάκων, είναι μείζον ζήτημα. Ιδίω σε ό,τι αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση. Και μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. λόγω του πολύ σημαντικού προβλήματος ε, της αντοχής ε, στα αντιβιωτικά. Μπορεί να είναι αποτελεσματική μια απαγόρευση. Είναι ένα θέμα που καλό θα ήταν να το θέσουμε στους ε, ειδικού για θέματα πληροφορικής. Εκεί θα υπήρχε πρόβλημα με την εποπτεία, άρα και με την επιβολή κυρώσεων ό,τι αφορά τώρα μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων, συμφωνώ, επί της αρχής τουλάχιστον, ωστόσο, θεωρώ ότι μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση θα ήταν η διάρθρωση ενδεχομένως ε, του οργανισμού φαρμάκων με καλύτερο τρόπο και αναφέρομαι στην έκθεση Τανέσκου εδώ. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία ενιαία πράξη για τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φάρμακων και όχι πολλές αναφορές ε, σε διάφορες νομοθετικές πράξεις. Επίσης, για τις παράλληλες εξαγωγές ή δοκιμή. Γίνονται κάποιες προτάσεις που νομίζω ότι πηγαίνουν λίγο μακριά. Υπάρχουν κάποιες καταχρηστικές πρακτικές, ε, είναι κάπως διαφλονικούμενα αυτά τα παράλληλα συστήματα, απαιτείται πολλή δουλειά και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της Επιτροπής και αυτή πρέπει να επιτελέσει το καθήκον της. Η ασφάλεια τώρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική τυχή ασφαλώς, πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και αποτελεί σαφή προτεραιότητα. Το ίδιο και τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι αρκετά. Το θέμα κυρίως είναι η ανάκληση και η διάθεση. Μίζον ζήτημα η διάθεση. Όλα τα κτηνιατρικά προϊόντα ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα να διατεθούν. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να ισχύσουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν για τα, για τα φάρμακα που προχωρίζονται για τον άνθρωπο και να υπάρξει σαφής κωδικοποίηση. Και στις εγκρίσεις, στα κυκλοφορίες των αντιβιωτικών θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς διαδικασίες, σαφώς ορισμένες. Τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται για ζώα, όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουν και μείζονες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει ένα σαφή συσχετισμό μεταξύ τη χρήση των άνθρωπων και τη χρήση στα ζώα και αυτή η διαδικασία, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ρυθμιστεί πάρα πολύ καλά και να οριστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε στην έγκριση του φαρμάκου είτε στην απόσυρση, στην απόρριψή του. Η έλεγχη επίση σε όλη την αλυσίδα της χονδρικής αλλά και της λιανικής πόλης είναι σημαντική. Και πρέπει να σας πω ότι έχω σκεφτεί ιδιαίτερα το θέμα της λιανικής πώλησης και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε έναν ανώτατο αριθμό ενίας άδεσης. Δεν ξέρω πώς χρειάζεται κάποιο κατόφυλλο, κάποια όρια, τον οποίο και μέσα σε μια συγκεκριμένη ποσότητα δεν μπορούν να εγκρίνονται περισσότερα φάρμακα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί βέβαια αυτό, αλλά νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η ομάδα των φιλελευθέρων και η κυρία Πάουλσεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκροστέτ γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις τροπολογίες της που αποσκοπούν σε τροποποιήσεις. Γιατί εδώ διευκρινίζομαι το περιεχόμενο του κανονισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για διευκρινήση και απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας αυτό στο νομοθετικό μας έργο. Συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουμε σαφή και κατανοητή νομοθεσία. Όχι μόνο εδώ, αλλά παντού, σε όλα τα νομοθετήματα. Τώρα, οι πωλήσει online στο διαδίκτυο αυτών των φαρμάκων. Έχω και μία τροπολογία για από την Επιτροπή Γεωργίας. Μία ερώτηση για την προφυλακτική θεραπεία που πρέπει να μην γίνεται, πρέπει να απαγορευτεί. Όταν μιλάμε για μικροβιακή αντοχή, ο, αν δούμε με τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι μας, είναι πολύ σημαντικός φορέας μόλυνσης αφού ζουν τόσο κοντά σε μας. Θα ήθελα λοιπόν όλα τα ζώα να συμπεριληφθούν στην απαγόρευση και όταν μιλάμε για περιβαλλοντικό αντίκτυπο εδώ μιλάμε για ανθιστάμενα βακτήρια και στο νερό και στα χωράφια και στο έδαφος που γίνονται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, ε, εδώ Τώρα αρχίζει η επιστήμη να ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα του προβλήματος. Γι' αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ σε αυτό το θέμα, παρόλο που δεν ξέρουμε ακριβώ πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά πρέπει να το προσέξουμε. Μία πρόταση λοιπόν, ε, να στηριχθούμε στην τροπολογία 65, δηλαδή να μην μιλήσουμε μόνο για τις υγειονομικές αρχές, αλλά και τις ε, αρχές αρμόδιες για το περιβάλλον και στα κράτη-μέλη και σε επίπεδο νοσιακό. Δηλαδή να ενημερώνονται για, με τον ίδιο τρόπο, να τους λέμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιβαλλοντικές αρχές. Επίσης είναι σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα από ό,τι προβλέπει σε ορισμένα σημεία του κανονισμός. Οι κτηνίατροι δεν πρέπει να πουλούν φάρμακα μάλλον να μην μπορούν να αποκομίζουν κέρδος από την πώληση αυτών των φαρμάκων. Αυτά πρέπει και στο μέλλον να χρειάζονται εξουσιοδότηση, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες εδώ. Τέλος. Ε, υπήρχε μια παράληψη στην πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή κανόνες για υπεύθυνη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Η πρόταση φαίνεται να εστιάζεται στα προϊόντα και όχι στα ζώα και τον άνθρωπο. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν ε, πιστεύω ότι είναι τελείως παράλογη. Δεν έχουμε προϊόντα που να μην έχουν ε, αντίκτυπο επίπτωση στα ζώα, στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και ειδικότερα δεν έχουμε φάρμακα γιατί αυτά παράγονται και χρησιμοποιούνται για να ασκήσουν κάποια επίδραση. Δεν μπορεί να μιλάμε σαν να είναι τεχνολογικά προϊόντα και όχι κομμάτι της ζωής μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και υπάρχουν και άλλες μικρολεπτομέρειες. Πάντως η συνεργασία μας είναι υποδειγματική. Η κυρία Γκροστέτ και εγώ είμαστε εδώ και πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και έτσι μπορούμε να πιστοποιήσουμε μεγάλη πρόοδο, γιατί μπορούμε να συνεργαζόμεθα σε πρακτικά θέματα. Αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ, ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συμφωνιών και συμβιβασμών. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο επόμενος ομιλητής από την ομάδα της αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Γκροστέτ, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά. Πολύ επικοδομητική επίσης, έλαβε υπόψη ευρύ το αριθμό σχολείων και επιθυμιών, ε, επέδειξε συμβιβαστικό πνεύμα και χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε ότι η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής θα τύχει προτεραιότητας ε, όπως και η εστίασή της στην προφυλακτική χρήση των φαρμάκων που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να τονίσουμε, κάτι που το ξεχνούν τα κράτη-μέλη, είναι η διάδοση πληροφοριών και η παροχή πληροφοριών, που είναι τόσο σημαντικό θέμα σήμερα. Καμιά φορά φαίνεται ότι το ξεχνάμε αυτό διότι θα πρέπει να καταδεικνύουμε στον κόσμο τους κινδύνους από τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα γενικότερα. Τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν πραγματικά χρειάζονται. Στην τροπολογία 81 ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και μάλιστα Σημειώνεται σε όλες τις τροπολογίες ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές αποστάσεις σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και την απόσταση στον ε, από τον πιο κοντινό κτηνίατρο. Αν υπάρξει κάποια νόσος, αν η γεωργική εκμετάλλευση είναι πολύ μακριά από το ιατρείο του κτηνιάτρου ή από το φαρμακείο σε εξαιρετικές τέλο πάντων περιπτώσεις η διάγνωση μπορεί να γίνεται και από το τηλέφωνο όταν τα ζώα είναι γνωστά. Τα γνωρίζει ο γιατρός. Και να μπορούν να συνταγογραφούνται και να απολούνται φάρμακα ιδιαίτερα στους αγρότες που έχουν πολλά βοηθή. Συχνά στη Φιλανδία τουλάχιστον συμβαίνει η απόσταση μεταξύ της εκμετάλλευσης και του φαρμακείου να είναι και 200 χιλιόμετρα. Οπότε η ιδέα να πάει ο κτηνίατρος στην αγροτική εκμετάλλευση και να συνταγογραφήσει ή να πάει ο αγρότης να τα πάρει, καλύπτοντας απόσταση 200 χιλιόμετρων, ε, είναι κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Τώρα για τα φάρμακα για τον άνθρωπο, αλλά και τα κτηνιατρικά φάρμακα, θα έλεγα ότι η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων παρουσιάζει προκλήσεις γιατί είναι μικρή. Η έρευνα ε, είναι αρκετά βραδία στα φάρμακα αυτά και αυτό, όπως είπα, δημιουργεί προκλήσεις. Όταν μιλάμε για εκτρεφόμενα ζώα ή κατοικίδια ή ζώα που χρησιμοποιούνται για σπόρ, οι ανάγκες είναι διαφορετικές και οι τρόποι φροντίδας των ζώων διαφέρουν. Οπότε ελπίζω οι κτηνίατροι να μην κατηγορηθούν ότι θέλουν να δώσουν στους ε, ε, πελάτες τους ε, ότι δεν θέλουν να δώσουν καλές υπηρεσίες και ότι προσφεύγουν σε φάρμακα να μην κατηγορηθούν ότι δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες όταν προσφεύγουν σε φάρμακα για τον άνθρωπο όταν δεν υπάρχει κτηνιατρικό φάρμακο. Είναι πολύ θετικό ότι τονίστηκε ιδιαίτερα η περιβαλλοντική προστασία. Και στο μέλλον να αποφεύγουμε ε, εκτιμήσεις και δράσεις που θα αποδυναμώσουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα το υδάτινο περιβάλλον. Νομίζω ότι με τη συνεργασία θα πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Να πω όμως ότι αυτό, αυτή η δέσμη νομοθετημάτων είναι πολύ δύσκολη. Αλλά παρόλα αυτά η κυρία Γκροστέτ έκανε καλή και επαγγελματική δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χόισλινγκ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ συμφωνώ σε πολλά σημεία. Θα προσθέσω όμως ορισμένα βασικά για την προβληματική. Το σχέδιο της Κομισιόν σε πολλά σημεία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη χορηγούνται διπλάσια κτηνιατρικά φάρμακα ε, από ό,τι για τον άνθρωπο. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται διορθωτικά με το σχέδιο της Κομισιόν, αυτό πρέπει να το πούμε. Όμως συμφωνώ με την προσέγγιση της κυρίας Γκροστέτ ότι πρώτα πρέπει να ορίσουμε την προφύλαξη και τη μεταφύλαξη. Η πρώτη πρέπει να απαγορεύεται. Αυτό δεν συζητείται καν. Η μεταφύλαξη είναι μια προσέγγιση. Τώρα, αν πηγαίνει ε, αρκετά ε, προς τη σωστή κατεύθυνση ορισμός πρέπει να το δούμε. Πρέπει να διατηρήσουμε υγιή ζώα και να αποφύγουμε ε, νόσους. Δεν μπορούμε να ε, διαχωρίζουμε εύκολα επίσης τα ζώα τα νοσούντα από τα υγιή. Και αυτό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει. Η απαγόρευση πολίσεων online, εδώ συμφωνούμε όλοι νομίζω, νομίζω ότι η κατάσταση αυτή θα ήταν ε, στο δινικές ανεξέλεγκτη, δεν μπορούμε να έχουμε εποπτεία, άρα συμφωνούμε στην απαγόρευση. Για ορισμένα προϊόντα όμως πρέπει να πω ιδιαίτερα με τις νέες εξελίξεις ε, φαρμάκων κτηνιατρικών έχουμε το πρόβλημα ότι ε, αναπτύσσεται κάτι στη βιομηχανία μόνο όταν μπορούν να εξασφαλιστούν κέρδη μέσα από μαζικές πωλήσει. Οπότε διευκολύνουμε τις ερευνητικές δυνατότητες και την ε, έγκριση ελπίζοντας ότι η βιομηχανία θα βγάλει στην αγορά φάρμακα. Είναι σωστό όμως αυτό ως προσέγγιση. Θα πρέπει ίσως να ε, δούμε και άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα γιατί τώρα τους διευκολύνουμε και ε, παρατείνουμε και τη διάρκεια ισχύωσης της εξουσιοδότησης, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι η μοναδική μας επιλογή. Ε, υπάρχουν κι άλλες. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, φαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων. Αυτό είναι ένα θέμα που πολύ σωστά απασχόλησε την κυρία Γκροστέτ. Δεν ξέρω αν πηγαίνει αρκετά μακριά γιατί υπάρχει και το θέμα ότι τα φάρμακα ε, μέχρι το 2003 δεν αξιολογούνταν ως προς και τώρα δεν προχωρούμε ε, αρκετά μακριά διότι μέσα από διάφορους, ε, διάφορες διάβλους φάνουν στο περιβάλλον τα αντιβιωτικά. Βρέθηκαν και στα υπόγεια είδα τα αντιβιωτικά στη Γερμανία και όλα αυτά κάπου καταλήγουν και έχουν επιπτώσεις σε, ε, με τρόπους που ακόμα δεν τους ε, έχουμε αρκετά ερευνήσει και πρέπει να ερευνήσουμε. Ένα άλλο θέμα που χρήζει καλύτερου ορισμού είναι το θέμα των εφεδρικών αντιβιωτικών. Ε, ιδιαίτερα στα ζώα χρησιμοποιούνται και αυτό είναι ένα μεγάλο κακό μακροπρόθεσμα δεν είναι αποδεκτό. Εδώ αφήσαμε ελευθερία στην Κομισιόν για να ορίσει το θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς. Υπάρχει ένας κατάλογος του ΠΟΗ για εφεδρικά αντιβιωτικά. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό ως κριτήριο ή αν θα προσθέσουμε κι άλλα που δεν θα τα επιτρέπουμε για κτηνιατρική χρήση, αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε διεξοδικότερα από ό,τι παρουσιάζεται στο σχέδιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπου θα μπορούσε κανείς να πάει πιο μακριά για να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν. Πάντως νομίζω ότι σε πολλά θέματα θα συμφωνήσουμε για κάτι καλύτερο που θα ανταποκρίνεται και στη σημερινή προβληματική. Και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία που θα οδηγήσει σε ικανοποιητικές ε, συμβιβαστικές λύσεις στο τέλος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η FTD. Ο κ. Πεντιτσίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε από μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν μας ικανοποιούσε και πάρα πολύ. Ήταν, δεν ήταν ισορροπημένη, ε, ισορροπημένη έτεινε προ τη φαρμακοβιομηχανία, κυρίως από τη γενική θέση της, στόχους της. Όταν θέλαμε να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα των κοινωτικών φαρμάκων και για τα μικρά είδη, όπως είναι οι μέλισσες, αυτό θεωρείται σαν αξίωμα, σχεδόν αναμφισβήτητο. Όμως χρειαζόταν μια θεολογική αντιμετώπιση. Και ε, έχουμε βολιαστεί το ΣΥΠΗΝ και έχουμε καταλάβει ότι ε, θέλουν να, να εκμεταλλευτούν οι, το, οι βιομηχανίες στον τομέα αυτό που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα. Θέλουμε την ευημερία των ζώων, αυτό είναι ο στόχο. Το να περάσουμε μαζική θεραπεία προ ατομικέ θεραπείε και εφαρμογή των σωστών πρακτικών σε αυτή την υγιεινή και σωστή διατροφή των ζώων, περνώντα από όλα αυτά προ την εκτατική κτηνοτροφία, ούτω ώστε τα ζεία να απολαμβάνουν ευρύτερο χώρο, καλύτερο περιβάλλον και να ζουν κανονικά. Διότι η υγεία των ζώων αντικατοπτρίζεται και στην ανθρώπινη υγεία Ανταυτού όμως είδαμε ότι ακολουθούσε αντίθετη κατεύθυνση η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόταση ηγήτρια όμως της κυρία Γκροστέτ έχει εισάγει διάφορες διορθώσει όσον αφορά την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την αρχική συζήτηση στηρίξαμε την απαγόρευση των πωλήσεων online συμφωνήσαμε με την απαγόρευση της προφυλακτικής χρήσης αυτών των προϊόντων. Ήμασταν αντίθετοι σε απεριόριστη ισχύ της έγκρισης και έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Πιστεύουμε δεν θα πρέπει να παρατείνουμε ε, την χρονική περίοδο προστασίας των μορίων. Για την ανθρώπινη χρήση η έρευνα των φαρμάκων ε, βασίζεται στην ε, σταδιακή αύξηση της ισχύω. Μπορούμε τη διάρκεια των αδειών να τη δώσουμε σε λιγότερες εταιρείες αν το κάνουμε αυτό θα διαχειρίζονται αυτές το κομμάτι της αγοράς. Οι λίγες επιχειρήσεις θα έχουν την άδεια. Πρέπει να το εξετάσουμε, το προσέξουμε. Και την χρήση off-label θα πρέπει να την προσέξουμε. Σε σύγκριση με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο στους ανθρώπους. Χρειάζεται πιο στενό πλαίσιο ρυθμιστικό για τη χρήση κάποιων φαρμάκων. που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ζώα. Off-label μόνο πρέπει να είναι έσχατη η λύση η χρήση των φαρμάκων αυτών. Όταν δεν υπάρχει απολύτως άλλη εναλλακτική. Όσον αφορά την εποπτεία των φαρμάκων, η προτείνηση γίνεται να υποστηρίξουμε την θέση της Κομισιόν. Αλλά έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Θέλουμε να μελετήσουμε την κατάσταση καλύτερα να προτείνουμε πιο αποτελεσματικέ λύσει δυνατόν. Σπυρίζουμε αυτό που είπε και η κυρία Πόλσον, ότι δεν θα πρέπει να πολλούν τα φάρμακα, να εκμεταλλεύονται προ την πώληση των φαρμάκων οι κτηνίατροι. Αυτό ήταν αρχικό στόχο. Συνολικά, εκτιμήσαμε τα μάλα το έργο τη ηγήτρια ε, και επιφυλασσόμεθα του να δώσουμε περαιτέρω ιδέες στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας. Η ε, κυρία Αγιούσο είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ και να επενέσω την κυρία Γκροστέτ για την πάρα πολύ καλή αυτή έκθεση με την οποία συμφωνώ θα σχεδόν στο 100%. Συμφωνώ ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία αυτή λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί επί του παρόντος όχι μόνο η διάθεση ε, των απορραντών, μιλώ για την εξάλληψή τους δηλαδή ε, και για ε, την, για ίσονο χρήση αλλά και τι γίνεται με τη μη εγκεκριμένη χρήση ή το διοικητικό βάρος που όλο αυτό συνεπάγεται και ιδίως η πρόθεση της απαραίτητης για αυτά τα φάρμακα αλλά και γενικότερα βέβαια της καινοτομίας ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων. Σίγουρα χρειαζόμαστε φάρμακα για τα διάφορα είδη και για τις παθολογίες, ιδίω για ίσονος σημασία και, ίσονος, και ίσονες χρήσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα ε, σπάνιδος φαρμάκων για τις πιο κοινέ νόσους, αλλά για τις πιο σπάνιες ή για τις ίσονες ε, χρήσεις έχουμε προβλήματα. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται εκεί πράγμα, φάρμακα που κανονικά προέρχονται για ανθρώπινη χρήση. Ό,τι αφορά το διοικητικό άκθος, ε, ε, συμφωνώ, αλλά μόνο όταν δεν έχουμε προσθέμενη αξία. Και πάντα πρέπει να αγγιόμαστε την ποιότητα, είναι το σημαντικότερο. Αλλά και την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια και την σωστή πληροφόρηση σε αυτούς τους τομείς δεν πρέπει να μειώσουμε το δικτικό βάρος. Επίσης θα πρέπει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η μικροβιακή αντοχή να το έχουμε υπόψη μας προς προς τη δημοσία υγεία δηλαδή, αλλά και την υπεύθυνη χρήση των αντιβιωτικών πρέπει να εξασφαλίσουμε όταν αυτά είναι απαραίτητα. Και θα πρέπει να γίνονται αξιολογήσεις, ε, εξέταση κόστους ωφέλους. Συμφωνώ λοιπόν με τις προτάσεις της κυρίας Γκροστέτ και σε ό,τι αφορά την ε, φάρμακο επαγρύπνηση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λίντς είναι επόμενος. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης Ευχαριστώ και για την καλή προκαταρκτική συνεργασία. με συντάκτες της νομοδότησης για τα φαρμακευτικά, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και νομίζω ότι θα καταλήξουμε, ότι καταλήξαμε μάλλον σε πολύ ε, καλές προτάσεις συνεκτικές γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους ίδιους ορισμούς και να υπάρχει σωστή εφαρμογή. Οι ορισμοί πρέπει να εξεταστούν καλύτερα, να γίνει διάκριση ε, προφύλαξης, μεταφύλαξης και θεραπευτικής χρήσης και είναι σωστό να προχωρήσουμε με πολύ περιοριστικό τρόπο εις ό,τι αφορά την προφυλακτική χρήση. Σημαντικός είναι ο κεντρικός ρόλος του κτηνιάτρου. Πρέπει να ενισχυθεί. Δεν νομίζω όπως η κυρία Πάουλτσεν, ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε το δικαίωμα διάθεσης φαρμάκων από το γιατρό. Ιδιαίτερα όταν δούμε, όταν, αν μειώσουμε το χρόνο συνταγογράφησης στις 7 μέρες ε, θα έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι μίλησαν και για τις πωλήσει από το διαδίκτυο. Νομίζω ότι σωστό είναι να απαγορευτεί αυτή και η επέκταση της διατήρησης των τεχνικών ε, εγγράφων ε, αντιμετωπίζεται σωστά από την κυρία Γκροστέτ. Μία πρόταση στο θέμα της ε, χρησιμοποίησης φαρμάκων για τον άνθρωπο στα ζώα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε αφενός να την περιορίσουμε και να είναι μόνο η έσχατη λύση και ίσως θα ήταν σωστό και απαραίτητο όταν χρησιμοποιούνται να δίνεται ε, έγκριση από την κτηνιατρική αρχή ούτως ώστε να μην αποφασίζει από μόνος του ο κτηνίατρος. Ίσως αυτό θα ήταν μια ε, λύση προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τα άλλα χαίρομαι για τη συνεργασία μας και νομίζω ότι είναι σημαντικό ιδιαίτερα να δούμε ολόκληρη τη δέσμη και στο τέλος να φτάσουμε σε συνεκτικές λύσεις. Αυτό είναι μια πρόκληση ε, γιατί σε αυτά τα θέματα η Επιτροπή Γεωργίας είναι αρμόδια επί της ουσίας και πρέπει να συντονιστούμε ούτω ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε ε, ίδιες λύσεις. Ευχαριστώ και αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ο επόμενος. Ευχαριστώ, ο Σπότς. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Πιστεύω, όπως και οι σκιώδεις εισηγητές, και εγώ θέλω να στηρίξω την όλη προσπάθεια, έχει στόχο τη βελτίωση της ε, προτάσεως και τίθενται αξιέπαινοι στόχοι. Καταρχάς, την αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βλέπουμε κατά πόσο η πρόταση κανονισμού ακολουθεί την κατεύθυνση της επίτευξης των τεθέντων στόχων. Νομίζω ότι η έκθεση της κυρίας Γκροστέτ ήδη καταβάλει μια προσπάθεια κάλυψης διαφόρων προβλημάτων που αρχική πρόταση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν συνέπεια την επιδείνωση της καταστάσεως νομίζω. Στην αρμόνιση δεν λαμβάνεται υπόψη η ευθύνη όσον αφορά την καταχώρηση των φαρμάκων. Δεν λαμβάνονται υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες κάποιων προϊόντων. Νομίζω ότι τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν καθορίζονται σαφώς. Και υπάρχει ο κίνδυνος μίας εναρμονήσεως όπου κάθε είδος φαρμάκου πρέπει να καλύπτει όλους τους στόχους. Και είναι δύσκολο να καλύπτονται όλα τα χαρακτηριστικά για όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Πρέπει να βασιστούμε και στις σωστές κτηνιατρικές πρακτικές. Όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, δεν καθορίζονται παρκώς οι διάφορες ευθύνες κατά τη διάθεση των φαρμάκων στην αγορά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφήνει πολύ ελεύθερο το πεδίο για κάποια φάρμακα που μπορούν να διατίθενται στην αγορά και αυτό εις βάρος της προστασίας των υγιών ζώων και της προστασίας της δημόσιας υγείας έχουν ασκηθεί πιέσεις από κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, φαίνεται αυτό, και θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Η πρόταση που υπευλήθη προσπαθεί να επιλύσει κάποια προβλήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν τους ελέγχους που δεν καλύπτονται. Θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα της αντιστάσεως στα αντιβιωτικά και αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε κοινή άποψη. Δεν πρόκειται περί πολιτικών ζητημάτων, αλλά δημοσίας υγείας είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Δεν είναι αποκλειστικά κτηνιατρικό, αλλά αφορά και τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση και την αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω να συνεργαστούμε και στο μέλλον επ' αυτού, διότι πρέπει να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να επαναξεταστεί λοιπόν η πρόταση αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Από κοινού θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Δεν είναι ασύνηθες αυτό, έτσι κάνουμε συνήθως με τις προτάσεις της Κομισιόν που τις φέρνουμε πιο κοντά στην πράξη. Τέσσερις διευκρινιστικές παρατηρήσεις συμπληρωματικές. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν χαίρομαι για την ε, ε, συμφωνία απαγόρευσης ε, σύντομα από το διαδίκτυο, γιατί αν το ε, απελευθερώσουμε δεν θα, θα χάσουμε τον έλεγχο και αυτό δεν είναι παραγωγικό. Δεύτερον, πρόκειται για το τι πρέπει και τι θα μπορεί να κάνει ο κτηνίατρος. Εδώ διαφέρουν οι απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν και σημαντικό θα ήταν ο κτηνίατρος να συνταγογραφεί και να δίνει τα φάρμακα, να τα χορηγεί. Η κυρία Πάουλσεν λέει ότι αυτό είναι πολύ ταπανηρό καμιά φορά. Εγώ ε, πιστεύω ότι πρέπει να είναι συνυπεύθυνο ο κτηνίατρος. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει διάλογος μεταξύ του κτηνοτρόφου και του ε, κτηνιάτρου. Την ε, διάγνωση την κάνει ο γιατρός, αλλά πρέπει να συνεννοηθούν για τη θεραπεία. Γιατί ε, αν γίνει λάθος η θεραπεία θα είναι υπεύθυνο ο κτηνίατρος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορεί και να χορηγεί τα φάρμακα. Τέλος να πω και ως ε, αγρότης Ε, όταν το κόστος ε, για τα φάρμακα είναι τόσο υψηλά όπως είναι σήμερα για τον ε, Γιωργό, κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως δεν πρέπει να είναι και υπερβολικά φθηνά. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση. Τρίτον, χρήση φαρμάκων για τον άνθρωπο και αντιβιωτικά. Εγώ θα ήθελα, αν έχουμε επακριβή ορισμό των εφεδρικών αντιβιωτικών, εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα ε, τέτοιο ορισμό και να απαγορεύσουμε άλλες χρήσεις. Ε, ο κ. Λίντς και η κυρία Πάουλσεν αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα των ε, κατοικιδίων που είναι ένας παράγωνα βεβαιότητας γιατί πολλές φορές επειδή αγαπάμε πολύ τα ζώα συντροφιάς μας τους δίνουμε φάρμακα που θα παίρναμε και οι ίδιοι ο κύριος Λίντς έκανε μια καλή πρόταση να φροντίσουμε τουλάχιστον ε, τα φάρμακα για τον άνθρωπο να περιορίζονται ε, με κριτήρια ασφαλείας. Αν ο κτηνίατρος όμως κάποια στιγμή καταλήξει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει φάρμακο για τον άνθρωπο στα ζώα, να παίρνει από μια ε, ανώτερη αρχή την άδεια. Ίσως αυτό θα μας εξασφάλιζε. Είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Γιατί πρέπει να προσέξουμε ε, και το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Τέλος, ε, άκουσα πολύ καλές προτάσεις από την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, τα στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα επίσης όχι μόνο στη Γεωργία να εφαρμόζονται αυτά, αλλά και στην ε, ιατρική γενικότερα. Είχαμε, ε, είχα συμμετάσχει σε ένα working dinner από όπου αποκόμισα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η ιατρική είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε στα πλαίσια της μικροβιακής αντοχής και δεύτερον, αν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση η γεωργία αλλά και η ιατρική για τον άνθρωπο τότε κάποια στιγμή η εποχή των αντιβιωτικών θα φτάσει στο τέλος της, γιατί θα έχει αυξηθεί το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Γκροστέτ για την έκθεση. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκροστέτ. Απέτησε πολλή δουλειά η έκθεση και το βλέπουμε αυτό. Θα επιμείνω επί των αντιβιωτικών. Και μετά στο πρόβλημα της καινοτομίας για τα αντιβιωτικά είδα τι γίνεται στη Δανία. Λέει ότι η Δανία μείωσε την συνταγογράφηση των ε, αντιβιωτικών υποχρεώντας τους νεάτρους να πουλούν το αντιβιωτικό. Κάθε φορά που ένας, ένας γεωργός χρησιμοποιεί το, το φάρμακο θα πρέπει να ενημερώνει τις αρχές. Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ των κτηνιάτρων και των φαρμακοποιών είναι σημαντικό. Και η λασιμότητα επίσης της χρήσης των αντιβιωτικών είναι σημαντικό. Στη Γαλλία θα είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, διότι οι κτηνίατροι έχουν ένα μέρος του μισθού τους που προέρχεται από την πώληση και των φαρμάκων. Αν θέλουν πραγματικά να επιτεθούμε στο πρόβλημα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα δύο. Το δεύτερο θέλω να πω είναι η καινοτομία. Έχω μία διαφωνία εδώ με εσά κυρία εισηγήτρια όσον αφορά την τροπολογία 42. Εκεί λέτε ότι θα πρέπει η περίοδος προστασίας της νέας τεχνικής τεκμηρίωσης για τα υφιστάμενα προϊόντα να είναι ετή. Για μένα αυτό είναι τροχοπέδι στον ανταγωνισμό και στην ενημέρωση. Αν θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε την καινοτομία δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιες προθεσμίες όπου δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την έρευνα για τα φάρμακα και αύξηση της έγκρισης και αυτό είναι τροχοπέδι για την καινοτομία. Λέτε ότι δεν είναι μεγάλη αγορά τα κτηνιατρικά φάρμακα, είναι όμως μια αγορά ε, της τάξης των 2 δις ευρώ δεν είναι κάτι αμελητήριο και το κέρδος των φαρμάκων συγκρίνεται με τα κέρδη για τα ανθρώπινα φάρμακα ανάμεσα στο 15 και 20%. Εκεί που συμφωνώ μαζί σας είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Νομίζω ότι η επισήμανση δεν αρκεί, χρειάζονται εκθέσεις υποχρεωτικές, τακτικά να υποβάλλονται και συμφωνώ μαζί σας. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος έχω κάποιο ερωτηματικό τι εννοείται με αυτή τη μονογραφή την περιβαλλοντική συναρτήσει των μορίων. Θα ψάχνουμε ποιες είναι οι συνέπειες των περιβάλλων. Ε, δίδονται τα φάρμακα στα ζώα. Το πρώτο στοιχείο που θα βρούμε την ε, επιρροή των φαρμάκων θα είναι και στο έδαφος και στο είδωρ. Θα πρέπει με τη μονογραφή να βλέπουμε τι γίνεται με τα ενεργά μόρια αλλά και τα πρόσθετες ουσίες. Πολύ συχνά δίδονται, βάζουν, προσθέτουμε ουσίες στο φάρμακο για να αυξήσουμε τις συνέπειες. Του Roundup. Θυμηθείτε τι έγινε με το μόριο της λικοζόδης που βάζαμε στο Roundup δεν είχε την ίδια δράση εκεί με το Roundup. Χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Θα πετύχουμε συμβαστικές λύσεις πιστεύω. Έτσι θα γίνεται καλή χρήση των φαρμάκων και καλή προστασία της ανθρώπινης υγείας παράλληλα. Διότι όσον αφορά ε, τα εφεδρικά αντιβιωτικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά και υπάρχει κάποιος κατάλογος όπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα εφεδρικά φάρμακα αντιβιωτικά μάλλον για τα ζώα και να χρησιμοποιούνται μόνο στους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια. Ε, καταρχάς, λέει κυρία Κουτλάντ, να τονίσω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που τόνισαν τη σημασία του θέματος. Πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα για το μέλλον. Αναφέρθηκε και η αντίσταση στα αντιβιωτικά και τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν επ' αυτού. Θέλω να πω ότι τελικά εδώ μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων. Και ήδη βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι απελπισμένος και όλο και περισσότερο στο μέλλον θα αυξάνονται τα προβλήματα. Και το έργο που επιτελείται είναι σημαντικότατο. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η σχέση μεταξύ της μη σωστής χρήσης της πενικυλίνης στα ζώα και ότι Έτσι δεν υπάρχει επαρκής προστασία των ζώων. Πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα, να προστατεύουμε την ευημερία των ζώων. Θα πρέπει να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες των, για τα ζώα. Αν προσφεύγουμε στα φάρμακα Ε, αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά φάρμακα και δεν θεραπεύονται σωστά τα ζώα, σημαίνει ότι δεν φροντίζουμε επαρκώς για τη σωστή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον κανονισμό και με τις τροπολογίες τελικά θα υπάρξει η σωστή προστασία και η διασύνδεση μεταξύ μαζικής χορηγήσεως φαρμάκων στα ζώα και των αντιβιωτικών με την αντίσταση κατά των ε, αντιβιωτικών απλωράς μικροβίων. Αν μεγαλώνουν τα ζώα σε κακές συνθήκες και δεν έχουν χώρο να ε, κινηθούν τα ζώα και επιτίθενται το ένα στο άλλο και τραυματίζονται όπως με τους χείρους. Όταν ασθενεί το ένα ζώο ασθενούν όλα τα ζώα και σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται μαζικά η πενικυλίνη δημιουργείται πρόβλημα. Είναι θέμα ευημερία των ζώων, προστασία της ευημερία των ζώων, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη συνταγογράφηση για τη χορήγηση των φαρμάκων από πλευρά των κτηνιάτρων. Δεν νομίζω ότι η σύγκρουση συμφερόντων του κτηνιάτρου είναι κάτι καλό. Να συνταγογραφεί το φάρμακο και μετά να έχει κέρδη από τη χορήγηση των φαρμάκων ο κτηνίατρος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι οι Γάλλοι κτηνίατροι θα πρέπει να εξηγήσουν πώς μπορούν να μειώσουν τη χορήγηση των φαρμάκων όταν εξαρτάται το κέρδος που βγάζουν από τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Επόμενη ομιλήτρια, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγροστέτ, χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε καταπιαστεί με αυτό το θέμα και θα συνεργαστούμε σίγουρα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι είμαι από την Ολλανδία και για πολλά χρόνια στην πολιτική όταν μιλάμε με, για τα γεωργικά αγροκτήματα, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εξετάζουμε τα στήματα αυτά και έχουμε, πρέπει να το πω, πετύχει αρκετά πολλά ήδη. Αν μιλάμε για κτηνιάτρους, κάποιες φορές ε, οι, του ΕΛΚ χρησιμοποιούν λίγο υποτιμητικά ε, τον όρο. Και το είδαμε και σε μια ακρόαση. Το ξέρετε ότι κάθε 15 μέρες πρέπει οι κτηνίατροι να επισκέπτονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να παρακολουθούν την κατάσταση, την καταχώρηση Και αν μιλάμε για αυτή τη μεγάλη μείωση, 45% και για κάποια που εργάζεται τόσο σκληρά, πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε και για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Θα πρέπει να δούμε και την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση. Θέλουμε να ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι και όχι μόνο, όλοι πρέπει να ενημερώνονται, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία και ένα ζήτημα που δεν αναφέρθηκε. Η συνέχεια, τι γίνεται, τι γίνεται, γίνεται μάλλον με τις ζωοτροφές. Στον Ολλανδία θέλουμε να θεσπίσουμε μέτρα παρακολούθηση για τι ζωοτροφέ. Ε, στα Μοσχάρια γίνεται ένα ε, σχετικό πρόγραμμα. Και αν θέλουμε να κάνουμε ελέγχου, αυτοί οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται διαφορετικά σε κάθε χώρα, αλλά με τον ίδιο τρόπο. Ίσως εμείς είμαστε πρωτοπόροι και μιλάμε για ένα 0,01% αλλά υπάρχουν Κάποιοι οποίοι δεν κάνουν τόσο αυστηρούς ελέγχους όσο κάνουμε εμείς, θα πρέπει λοιπόν να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι με πολύ αυστηρό τρόπο. Ακούμε τα νούμερα, πρέπει να δούμε και το βάρος απόδειξης. Από κοινού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Την τελευταία φορά είχαμε συζητήσει τον τομέα των πουλερικών. Εγώ μελέτησα τις πληροφορίες Είχαμε ένα καθηγητή από την Ουτρέχτη, τον Ιωάννη Φούνκε, που μας έκανε μια παρουσίαση. Νομίζω ότι η πρότασή σας μπορεί να είναι ικανοποιητική για τον τομέα των πουλερικών. Πρόεδρος. Κυρία Όκεν, τους Πρασίνους, τελευταίο μιλητρία. Ευχαριστώ. Να κάνω ένα επιπλέον σχόλιο κι εγώ και έχει να κάνει με τις τελευταίες εξέλιξεις. Η Δανία έχει ίσως από τα καλύτερα ιστορικά στο τομέα του ελέγχου των ε, κτηνιατρικών φαρμάκων. Είμαστε από τους, θα έλεγα, οι Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Στο πρωτοσέλιδο της πολιτικής μιας, μιας πολύ σημαντικής εφημερίδας λέει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν ε, σε μια οικογένεια που ασχολείται με την εκτροφή χείρων, έχουν προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς, δεν τους δέχονται ε, και νοσοκομεία και παιδική σταθμή κτλ. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των, ε, της σύγκρουσης συμφερόντων ή των διαφορετικών συμφερόντων. Δεν μιλάμε βέβαια για την ηθική και τη διοντολογία γιατρού και την ιάτρου εδώ. Κάποιοι που μπορεί να έχουν μετοχές ή να εξαρτώνται από τη φαρμακοβιομηχανία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όλοι αυτοί και ηθικοί και πιστοί αλλά τη σύγκρουση συμφέροντων πρέπει να τα αποφύγουμε. Και αυτό πρέπει να είναι μια αρχή και για τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα φάρμακα που προορίζονται για τα ζώα. Θα πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια και να απαγορεύεται να υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση, οποιαδήποτε σχέση γιατρών, κτηνιάτρων με φαρμακοβιομηχανίες και τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Έχουμε κάποιους εκπροσώπους ε, του κελπνού, του αντίστοιχου. And I would pass the floor. Και του οργανισμού φαρμάκων. Ποιος θέλει το λόγο. Κανείς. Προχωράμε λοιπόν και δίνω το λόγο στον κύριο Ρης, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στη σημαντική αυτή συζήτηση. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια βασικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν και από την έκθεση και από την σημερινή συζήτηση. Ο πρώτος σημαντικός τομέας είναι οι ορισμοί που χρησιμοποιούμε στην πρότασή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαρά να βοηθήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν επί των ορισμών. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ε, καταρχήν δεν μπορεί να υπάρξει επικαιροποίηση των ορισμών με κατεξουσιοδότηση πράξη. Άπας και υπάρχει ένας ορισμός, ο αντίκτυπός του παραμένει για χρόνια και για δεκαετίες, που του λεχθέντος, όταν ε, επεξεργαστήκαμε και εμείς την πρόταση, προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε και να ορίσουμε καλύτερα κάποια ζητήματα, χωρίς αυτό να μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο. On other point is the... Ένα άλλο σημείο είναι πρωτοβουλίες για καινοτομία. άκρος πολύπλοκο το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι προτινόμενες τροπολογίες θεωρούν ότι οι συμβασμοί πρέπει να είναι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες, ιδίως μιλώντας για ίσονα είδη στην πρόταση Κομισιόν. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να συνεπάρξει αυτό με την πρόταση που κάνουμε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια για να υπάρχει συνεκτικότητα, συνέπεια στο κείμενο. Επίσης, θα θέλαμε και τη συζήτηση στο το, τομέα αυτό να την διευρύνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μικροβιακή αντοχή, είναι σημαντικό. Είναι προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καλωσορίζουμε τις προτάσεις του κειμένου για ενίσχυση αυτού του συστήματος, αλλά θα πρέπει να δούμε και ότι υπάρχουν και κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην πρόταση. Και θα πρέπει να δούμε ολιστικά πώς μπορεί όλο το σύστημα αυτό να λειτουργήσει. Είναι σημαντικό. Να μπορούν να λειτουργήσουν όλες αυτές οι προτάσεις για να μην υπάρχουν καταχρήσεις των αντιμικροβιακών φαρμάκων ε, για τη θεραπευτική αγωγή των ζώων σε ό,τι αφορά την παράλληλη εισαγωγή και την παράλληλη διανομή. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η χρήση φαρμάκων εκτός ενδείξεων προβλέπεται στο 115 και 116 Αυτό είναι διαφορετικό από τη λεγόμενη παράλληλη εισαγωγή και παράλληλη διανομή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις παράλληλες διότι δεν θεωρήθηκε ότι ήταν σκόπιμο από τη στιγμή που υπάρχουν οι εθνικοί κανόνες. Αυτό λοιπόν προς διευκρίνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χονδρική ε, πώληση, διανομή, είναι καλή ιδέα. Θεωρούμε ότι οι νέε διατάξεις δεδομένων των προδιαγραφών για τον κτηνιατρικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν. Έχουμε καλά παραδείγματα από τα φάρμακα που προέρχονται για ανθρώπινη χρήση. Εκεί καταφέραμε να δημοσιεύσουμε το 2013 κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές διανομής. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε τις διατάξεις αυτές και στο τελικό κείμενο. Σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σίγουρη ως προς το τι πρέπει να καλύπτεται υπό την έννοια της εναρμόνισης των συνθήκων χρήσης έναντι της εναρμόνισης των, της περίληψης των χαρακτηριστικών προϊόντων. Ποιο μέρος περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντων δεν θεωρεί η συγκήτρια ότι δεν πρέπει να εναρμονιστεί. Βέβαια αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι άκρος πολύπλοκο το θέμα αυτό σίγουρα πάντα η εναρμόνιση είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, έρχομαι στη φαρμακοεπαγρύπνηση και σημειώνω τις προτάσεις. Ο στόχος μείωσης των διοικητικών βαρών σε σχέση με τη φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένας λόγος. Έχουμε και την έννοια ε, της ε, μεγαλύτερης συνέπειας. Σίγουρα ο συνδυασμό των δύο συστημάτων, δηλαδή να έχουμε και την αντιμετώπιση και το PCR και του ε, κινδύνου, ανείχνευση των κινδύνων, ίσω να είναι πράγματι ε, να συνεπάγεται αύξηση των δικαιωτικών βάρων. Θα πρέπει να το δούμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά την ε, τίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στόχος μας είναι να μην επαναλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές μελέτες όταν αυτό δεν αιτιολογείται επιστημονικά αλλά είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε ρεαλιστική πρόταση να την εξετάσουμε. Αν δηλαδή είναι εφικτό το να έχουμε ένα σύστημα μονογραφίας. Θα δούμε. Ίσως χρειαστεί να μας βοηθήσει εδώ περισσότερο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου που έχει ήδη κάποια εμπειρία. Ίσως το τελευταίο τώρα σχολείο μου επισήμανση να επαναλάβω ότι είμαστε υπέρμαχοι της απλούστερης αλλά και πιο αποτελεσματικής δυνατής επισήμασης. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο διοικητικό βάρος η σωστή επισήμαση. Και τέλος, ένα σχόλιο για τους κτηνιάτρους, γιατί το ανέφεραν αρκετοί βουλευτές. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή δεν έχει να κάνει με τη ρύθμιση κάποιου επαγγέλματος αλλά για τη ρύθμιση ιατρικών προϊόντων. Και σίγουρα ιατρή πρέπει να παραμένουν στο δυνατόν πιο ανεξάρτητοι επαγγελματίε, προσιλωμένοι στους βασικούς στόχους αυτής της πρότασης, μεταξύ των οποίων είναι και η μειωμένη χρήση αντιβιωτικών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στον τομέα αυτό. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Α, και τώρα η συγγήτρια έχει και πάλι το λόγο. Κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα ευχαριστήσω καταρχάς πραγματικά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι παρενέβησαν. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε το σύνολο των προσανατολισμών της εκθέσεως. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι μαζί θα καταλήξουμε στην επεξεργασία ενός κανονισμού αποτελεσματικού και χρήσιμου που θα επιτρέψει την επίλυση κάποιων προβλημάτων γνωστών σε μας σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι σημείωσα τα όσα μου είπατε και θα εξετάσω τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε και θα προσπαθήσουμε πράγματι να κινηθούμε μαζί ούτως ώστε να έχουμε έναν πολύ καλό κανονισμό θα σηματοδοτήσω εντάχει κάποια ζητήματα που εφήγησαν. Δεν μπορώ να επισέλθω στις λεπτομέρειες. Γνωρίζω ότι ο κ. Θανασέσκου, σκιώδης εισηγητής, συμφωνεί με τις προτάσεις αυτών των φαρμάκων που δεν χρησιμοποιούνται, για την χνηλάτιση αυτών, για την κεντρική συγκέντρωση των πληροφοριών θα πρέπει να θαρρυθεί η κεντρική διαχείριση. Είναι και αντικείμενο των τροπολογιών 1, 44 και 46 που υπέβαλα, αλλά ο κατακαιρματισμός της αγοράς καθιστά αναγκαία τη διαδικασία την αποκεντρωμένη, ακόμα και αν θα ήταν ευκταίο να έχουμε κεντρική διαδικασία, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη όσον αφορά τη συνταγογράφηση και την πώληση Πεσιώνω στο 81 πεσιώνω τη συνταγογράφηση υπάρχουν κάποιες διαγνώσεις κτηνιατρικές που θα πρέπει να δίδονται ε, μετά την εξέταση και θα πρέπει να ακολουθείται και ένα πρωτόκολλο θεραπείας το θέμα της αποσύνδεσης τέθη υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές όμως στα διάφορα κράτη-μέλη Στι σκανδιναβικέ χώρε έχουν προχωρήσει περισσότερο σε βάση συνταγογράφηση και πόσε κτηνιάτρους. Υπάρχουν πολύ καλέ πρακτικέ που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να διαδοθούν. Σήμερα όμω, το θεωρώ δυσχερέστατο, ανέφικτο να γίνει αυτό αντιμετωπίζουν προβλήματα οι γεωργοί και κτηνίατροι κάποιοι που είναι απομονωμένοι, που απέχουν πολύ από τα φαρμακεία. Χρειάζονται την πώληση από τον κτηνίατρο. Θα προσπαθήσω να το ρυθμίσω αυτό συγκεκριμένα στον κανονισμό, να μην υπάρχει κατάχρηση για τον καθορισμό της ε, προφύλαξης τα κατοικίδια ζώα να συμπεριλαμβάνονται στην απαγόρευση επικυρία Πόλσον και εγώ λέω ότι έχει δίκιο γιατί όχι και υπάρχει και, ένα σχετική, σχετική τροπολογία 97 όσον αφορά την ε, εκ αντιμετώπιση είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε την μόλυνση όλων των ζώων ε, μιας εκμετάλλευσης. Λένε ότι πρέπει να απομονώνεται το άρρωστο ζώο εξαρτάται από το ποιο ζώο ε, τρέφεται. Ας πούμε στα πουλερικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Στα βοηδή ίσως είναι πιο εύκολο απομονωθεί το στο ζώο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα προς επίλυση. Ο κύριος Άουσλινγκ προτείνει να απομονώνονται τα ασθενή ζώα. Σε κάποιες περιπτώσεις λέω ναι, αλλά ίσως να κοστίζει και στους κτηνιάτους κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όσον αφορά το περιβάλλον, Όλοι θέλετε να προστατεύετε το περιβάλλον, το κατανοώ, πολύ αναφερθήκατε σε αυτό, συμφωνώ μαζί σας. Πρότεινα να υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής μονογραφίας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική μονογραφία θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις, διότι μου ζητήθηκε, όπως από την κυρία Ριβαζή. Αξιολογούμε τις ενεργούς του εν πρώτης και εν συνεχεία αξιολογούμε τον αντίκτυπο του προϊόντος σε σχετισμό με τα διάφορα και τα διάφορα συστατικά του φαρμάκου. Μπορούμε να κάνουμε σε δύο στάδια αξιολόγηση. Μονογραφία για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο μιας ενεργού ουσίας που υπάρχει στο προϊόν και εν συνεχεία μια αξιολόγηση του αντικτύπου κατά προϊόν που θα είναι κάτι πιο εύκολο, διότι ο αντίκτυπος ενεργού ουσίας ήδη θα έχει αξιολογηθεί. Πράγματι υπάρχουν ε, πρακτικές ε, δυσκολίες, είναι σαφές αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει λεπτομερή έκθεση που θα επιτρέπει τον καθορισμό των πρακτικών λεπτομεριών. Όσον αφορά τον κατάλογο των αντιβιωτικών, των κυσίμων εφεδρικών, Τη τροπολογία 38 και 39 τη δικέ μου λέω να υπάρχουν κριτήρια για, τον, για την κατάρτιση των καταλόγων αυτών μετά από συστάσεις τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Σίγουρα υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά την κατάρτιση των καταλόγων. Εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μα πει, να μα καθαρίσει κάπω τι εννοεί. Για τα κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου και των καταλόγων. Θα υπήρχαν πολλά άλλα που θα μπορούσα να αναφέρω, που εθίγησαν. Νομίζω ότι δεν μπορώ να μακρηγορήσω τώρα, αναφερόμενοι σε όλα όσα εθίγησαν. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, διότι είδα ότι ο κανονισμός αυτός και η έκθεση δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω στους συναδέλφους, τους επιφορτισμένους με τα φάρμακα αυτά και τα τρόφιμα που περιέχουν φάρμακα ότι χρειάζεται εναρμόνιση, συνοχή μεταξύ των δύο κειμένων. Ήδη συνεργαστήκαμε. Θα συνεχιστεί αυτό. Θέλω να σας πω, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για όλα όσα είπατε. Θα συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι ένα καλό κείμενο. Χάρη σε όλους σας. Είμαι ανοιχτή στις συστάσεις σας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη συνεργασία που θα συνεχιστεί. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 15 Ιουνίου, 4 το απόγευμα. Ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες. 15 και 16 Ιουλίου. Η ακριβή ημερομηνία θα καθοριστεί αργότερα. Αναμένει ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 22 Σεπτεμβρίου μετά τις θερινές διακόπες. Δεν έχουμε πληροφορίες τώρα όσον αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Εξαρτάται και από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους, τη συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, τους κοιόδης και τα μέλη. Και προχωράμε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Τροποποίηση του κανονισμού 726 κάθετος 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης αδείας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Καταρχάς, το λόγο έχει ο συγγητής, ο κ. Τσίπριαν Θανασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όπως είπαμε και πριν εδώ στην Επιτροπή, θεωρώ ότι είναι θετικό το βήμα της Κομισιόν που προτείνει αποσύνδεση της έγκρισης εξουσιοδότησης κτηνιατρικών φαρμάκων από Κίνα για τον άνθρωπο για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του κτηνιατρικού τομέα. Επίσης σύμφωνο με την ευθυγράμμιση προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όμως όπως βλέπετε από το σχέδιο έκθεσής μου, εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που χρήζουν βελτίωση. Διαφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν για την δομή και το ύψος των τελών δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκτελεστική πράξη για τη διάρθρωση και το ύψος των τελών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στον καθορισμό των τελών του οργανισμού μέσα από την συνήθι νομοθετική διαδικασία. Προτείνω και κάποιες τροπολογίες για διευκρίνηση και ε, ενημέρωση των τελών που ισχύουν ε, για, ε, που πρέπει να καταλαμβάνονται στον οργανισμό με βάση τα άρθρα 563 που ορίζουν τις διάφορες πηγές ε, εσόδων για τον οργανισμό από κτηνιατρικά και άλλα φάρμακα για τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών τύπων εσόδων που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό του οργανισμού. Άλλες τροπολογίες ε, αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι ο κανονισμός θα ευθυγραμμίζεται με τον οικονομικό, δημοσιονομικό κανονισμό ώστε να ε, διευκολύνεται πρόσβαση και σε άλλες πηγές ε, χρηματοδότησης. Ευθυγράμμιση με άλλες πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα ή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, δηλαδή θα υποστηρίζουν τις εργασίες με αντικείμενο τα προγράμματα δημόσιας υγείας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, ρύθμιση στον κανονισμό του ρόλου του αίμα στη χορήγηση άδειας λειτουργίας και την εποπτεία των κτηνιατρικών προϊόντων. Ε, επίσης, ε, ο ισχύων κανονισμός 297 του 95 για το γενικό καθεστώς θελών του αίμα και το ε, κανονισμού 658 του 2014 για τα τέλη φάρμακο επαγρύπνησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη νομική βάση μέχρι την αναθεώρηση του κανονισμού 297 ή έως ότου θεσπιστούν και τεθούν σε εφαρμογή άλλες διατάξεις σχετικά με τα τέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα στους σκιώδεις. Η πρώτη ομιλία είναι από το ΕΛΚΑ και η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδη ηγήτρια. Ο κύριος Σεριός συνάδελφός μου είναι, αλλά απουσιάζει σήμερα και μου ζήτησε να μιλήσω στη θέση του και με τα χαρά στο κάνω. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των κειμένων αυτών που αφορούν ένα κοινό θέμα. Ο συνάδελφός μου, κύριο Συριό, θέλει πραγματικά να συγχαρεί όπως και εγώ τον κύριο Θανασέσκου για την έκθεσή του. Συμφωνεί απολύτως με τη βάση της εκθέσεως και θέλει να τον ευχαριστήσει για την άριστη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ τους. Ο κύριος Συριό ανησυχεί, όπως και ο για δύο συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο, αφορά τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων για τις αστηριότητες στον κτηνιατρικό τομέα. Σύμφωνα την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά θα πρέπει να καθορίζονται από εκτελεστική πράξη και ο κύριος Συριώπους και ο συγητής προτιμούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νέα νομοθετική πράξη από αυτού. Δεύτερο σημείο αφορά τη διάρκεια της ανάθεσης εξουσιών που χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή είναι αόριστη στην αρχική πρόταση, διάρκεια. Ο εισηγητής προτείνει περιορισμό σε πενταετία και ο κ. Συριό θα ήθελε να κινηθεί προς την της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνεί επί περίοδου περιορισμένης, αλλά θα θεωρούσε ότι αυτή η περίοδος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της πενταετίας είναι μια απόχρωση σχετικά με τη θέση του συγητού. Αυτά είναι τα βασικά σχόλια του σκιώδου συγητού του, που θα έκανε ο κ. Σιριό εκ μέρους του ΕΛΚΑ ήταν παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής από την ECR, ο κ. Πιεχάινεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή Εκτιμώ την όλη προσπάθεια, τον ζήλο, το έργο, προσωπικά και εξ ονόματος της ομάδας μου, της ECR, στηρίζω την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογική η προσέγγιση σε μια νομική πράξη Συμφωνώ επίσης με την αποσύνδεση, με αυτή την αρχή της αποσύνδεσης αδειών κυκλοφορίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα από τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Αλλά υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της μείωσης των προτύπων, γιατί κάποια γενώσιμα είναι παλιά. Αυτά δεν προκαλούν πρόβλημα. Όμως, στα πλαίσια της καινοτομίας μπορεί να πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα και αντιβιωτικά σε περίπτωση καινοτόμων προϊόντων και αντιβιωτικών οι διαδικασίες πρέπει να είναι συμβατές με εκείνες που αφορούν στον άνθρωπο. Συμφωνώ με τη δομή των τελών, τη διάρθρωση των τελών, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να γίνεται ρυθμίση από κοινού για τους αντίστοιχους οργανισμούς από τα κράτη-μέλη και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει συνένεση που θα είναι αποδεκτή και από τη βιομηχανία και από τις κυβερνήσεις μας γιατί Βέβαια, η βιομηχανία πρέπει να επομιστεί ένα σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα, όπου τα ποσά για τα οποία μιλάμε μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την διαφάνεια. Αναφέρομαι στο άρθρο 67 στο τμήμα 3 που έχει να κάνει με τα έσοδα του οργανισμού. Στο σημείο 3 αναφέρονται άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός. Τι σημαίνει αυτό, τι είδους υπηρεσίες είναι αυτές. Μπορεί η ερμηνεία εδώ να μην είναι εύκολη, οπότε μπορεί εδώ να έχουμε να αντιμετωπίσουμε υψηλό κόστος για τον παρασκευαστεί. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Στην προηγούμενη παρέμβασή μου, όταν μιλούσαμε για την έκθεση Γκροστέτ, μίλησα για βάσεις δεδομένων και περιλήψεις χαρακτηριστικών φαρμάκων. Ε, επισημάνσεις, φυλάδια, ενημερωτικά. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε μια αποσύνδεση ή διαχωρισμό που θα είναι σημαντικός μεταξύ των φαρμάκων για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αυτό θα είναι πιο εύκολο και για τους ασθενείς και τους καταναλωτές και τους κτηνιάτρους και τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Τώρα, επανέρχομαι στα τέλη τα οποία πρέπει να προσαρμόζονται προς τις εξελίξεις στη βιομηχανία. Εγώ μίλησα πολύ με εκπροσώπους του κλάδου της βιομηχανίας και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα παρασκευάζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε ο κλάδος να μπορεί να δαπανά σημαντικό ε, ποσό των διαθέσιμων κονδυλίων στην καινοτομία, ούτως ώστε να είναι καλά τα προϊόντα. Άρα τα τέλη πρέπει να είναι λογικά σε αποδεκτά επίπεδα για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Και να έχουν περιθώριο ελιγμών Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις τροπολογίες, ε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε και τον κύριο Τανασέσκου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή εδώ είναι μάλλον τεχνικός ο φάκελος συνδεδεμένος με τον προηγούμενο εν προκειμένου πρόκειται για την αποσύνδεση των αδειών κυκλοφορίας για κτηνιατρικά και μη φάρμακα αυτό είναι όχι μόνο λογικό για τον τομέα και συμφωνώ να βγάλουμε τα κτηνιατρικά από το κείμενο, αλλά είναι και προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε όλα είναι πολύ σωστά. Ορθότατα και συμφωνώ με τον εισηγητή σε όλα σχεδόν όσα έκανε. Για τα τέλη, η Κομισιόν προτείνει να έχουμε κανονισμό του Συμβουλίου και όπως ο εισηγητής πιστεύω ότι εν προκειμένου πρέπει να υπάρξει συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ δικαιολογημένο και έχει πολύ νόημα. Ε, δεν θα πω ε, περισσότερα, αυτά είναι τα βασικά άλλωστε τα θέματα της έκθεσης και περιμένω με ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Χόισλινγκ, ο Σκιώδης από τους Πρασίνους. Και εγώ ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή, συμφωνούμε σε πολλά, είναι τεχνικός, τεχνική έκθεση, αλλά δεν σημαίνει ότι ε, χρειάζεται λιγότερη δουλειά. Μια παρατήρηση για το σύστημα των μονογραφιών. Θα θέλαμε ενημέρωση για τις δραστικές ουσίες στα κτηνιατρικά φάρμακα να συλλέγεται σε κεντρικό επίπεδο και να διατίθεται στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολύνονται ε, στην συλλογή αυτών των δεδομένων. Η βάση δεδομένων για τις δραστικές ουσίες θα πρέπει να δημιουργηθεί και θα πρέπει να εξασφαλίζεται δωρεάν πρόσβαση από όλου και σε τακτά διαστήματα να ενημερώνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να ε, δείξουμε στην κοινή γνώμη μια αγορά που χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες και ανταλλαγή πληροφοριών που θα κοινοποιούνται και στην κοινή γνώμη ευρύτερα. Αυτό είναι σημαντικό να το συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόισλινγκ και τώρα από ο κύριος Πεντιτσίνη από την ομάδα FTP. FTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς εκτιμούμε την πρόταση του εισηγητού του κ. Τανασέσκου για τις γενικές γραμμές που ακολουθεί. Εφηγραμμιζόμαστε με την αρχή και με όλες τις προτάσεις που είναι υπέρ νομικών δίσων που ε, αφορούν πλήρη εμπλοκή το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να πρόταση να επιτρέψει στο Ευρωκοινοβούλιο τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά την καταπολέμηση των προβλημάτων και των θέσπιση των διαδικασιών για την αδειοδότηση. Η ξεζώτηση πράξης ε, καλύπτουν τι μη ουσιαστικέ πτυχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει ε, ε, πράξεις νομικού περιεχομένου. Να θυμηθούμε ότι εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι αυτές οι εν πράξεις τι κάνουν. Και θα ζητούμε ανάκληση ε, αν είναι αντίθετε με τη συνθήκη. Και στην Ολομέλεια θα δούμε κατά πόσο οι κατοξιδότητες στην πράξη παραβιάζουν τις βασικές πράξεις. Θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις αφού έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε ενδελεχέστερα την όλη πρόταση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πεντιτσίνη. Και τώρα Ο κύριος Ρης, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μήπως μπορεί να συμβάλλει στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όσα υπόθηκαν. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ε, σχέση μεταξύ των νομοθετικών πράξεων και πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι σωστές διασύνδεσεις Πρέπει να βρούμε καλύτερο τρόπο να το εξηγήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Σημαντικό θέμα αναφέρει η έκθεση. Τη διάθρωση των διαφόρων στοιχείων. Και τι γίνεται σε σχέση με την απόφαση του ΔΕΚ του 2012 για τις εξουσίες που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό των τελών. Ελέγξαμε ποιοι φορείς για ποιους φορείς καθορίζει τα τέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την υπηρεσία των χημικών ουσιών, αυτό έχει γίνει το 2013, υπηρεσία ανοτομία το 2014. και την αρχή για τους τίτλους και τις χρηματοστατικές υπηρεσίες το 2012. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό στηρίζω τη δική μας θέση. Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 70α. Δεν αναστέλλεται το, το παρόν καθεστώς τελών, αλλά καθορίζεται η βάση των μελλοντικών τελών, ίσως το άρθρο 70α. Ίσως η αναφορά αυτή θα έπρεπε να μπει σε τελικέ σκέψει. και οι ταξινομήσεις των εσόδων τη υπηρεσία συζητούνται. Θα βοηθήσει το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σωστή διατύπωση για τα δύο άθρα που θα αντικατοπτρίζουν του πόρου τη υπηρεσία και τη διαδικασίες απαλλαγή, χωρί να υπονομεύουμε την εντολή τη υπηρεσία και το νομικό πλαίσιο εντό του οποίου κινείται. Τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή κύριο Τανασέσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιμένω τα σχόλια και τις προτάσεις των συναδέλφων μέχρι τη λήξη της προθεσμής για την κατάθεση τροπολογιών και έχω την εντύπωση ότι κάναμε μια καλή αρχή θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους και αυτό πιστεύω θα οδηγήσει σε μια καλή έκθεση. Και πάλι ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και παραμένω στη διάθεσή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν ναι, στη συζήτηση. Να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 15 Ιουνίου 4 το μεσημέρι. 15 Ιουνίου παραλαμβάνω 4 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή ΕΝΒΗ θα ψηφίσουμε στις 22 Σεπτεμβρίου. Δεν σας εκπλήσει. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε για το προηγούμενο θέμα μας. Και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ημερομηνία. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Μείωση των εκπομπών ρήπων από οδικά οχήματα.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 Όπως είπε ο πρόεδρος, ο συνάδελφος Άλμπερτ Ντες δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και με παρακάλεσε γι' αυτό να παρουσιάσω την έκθεσή του που είναι μάλλον τεχνική έκθεση και παρακαλώ την κατανόησή σας. Ε, θα διαβάσω τις ε, προτάσεις του. Η πρόταση αποτελείται από ετερογενή μέτρα που στόχο έχουν την ανθρώπινη υγεία απέναντι στις εκπομπές της λαβερές. Τα μέτρα αυτά αφορούν τον καθορισμό συγκεκριμένων οριακών τιμών για το διοξίδιο του αζότου στα πλαίσια των εκπομπών ε, οξυδίων του αζότου. Δεύτερον, η μη χρήση των ε, τιμών των οριακών για την αμμονία, κατάργηση του ορίου δηλαδή, ε, επίσης ε, ε, να έχουμε μία τροποποίηση των ορίων εκπομπών κίνησης, ψυχρής εκκίνησης από τα πρότυπα τα προηγούμενα, ένα μέτρο προσαρμογής των συνολικών εκπομπών υδρογων ανθράκων για την εισαγωγή φυσικού αερίου, να υπάρχει δυνατότητα να προσθεθεί το μεθάνιο και να υπάρξει δυνατότητα εκπαίδευση, ε, επέκτασης από 2.840 στις 5.000 χιλιόγραμμα. υπάρχουν και άλλα μέτρα πιο τεχνικού ρυθμιστικού χαρακτήρα, αφορούν περιπτώσεις όπου προτείνεται η ευθυγράμμιση εκτελεστικών εξουσιών τα σημερινά νομοθετικά κείμενα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και κάποιες ε, νέες εκτελεστικές εξουσίες που θα λειτουργήσουν ως μέσο εφαρμογής μερικών από τα νέα προτινόμενα μέτρα. Ε, καταρχήν κάθε μέτρο που βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ευπρόσδεκτο, ιδίω όταν καταφέρει να εξισορροπεί αποτελεσματικά δαπάνες και αποτελέσματα με τη μορφή βιωσιμότερων πόλεων, όπου συγκεντρώνονται πολλοί. Ε, κάτοικοι. Ε, θα πρέπει επίσης να ε, μειώσουμε εκπομπές υπέρ της ανθρώπινης υγείας, να έχουμε και χαμηλότερες δαπάνες βέβαια για την υγεία. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να επιβάλλονται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων μέτρα που τους δημιουργούν τις ανάλογες επιβαρύνσεις. Ε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο κλάδος εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προσπαθεί να αποτινάξει τις συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και ότι οποιασδήποτε πρόσφατες δαπάνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν. Ο εισηγητή επιθυμεί λοιπόν να επισημάνει ορισμένε συγκεκριμένε παραμέτρου τη πρόταση τη Επιτροπή και των προτινόμενων τροπολογιών. Δεν θεωρεί ότι το μεθάνιο ε, ε, δεν θεωρεί ότι είναι ρηπογόνο ε, αέριο το μεθάνιο από μόνο του και δεν συνιστά απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Τα οχήματα φυσικού αερίου εκπέμπουν όμως περίπου 25% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από τα οχήματα που καίνε πετρέλαιο. Και τώρα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το μερίδιο αγοράς που θα καταλάβουν στο μέλλον τα ε, οχήματα με αέριο. Αυτά τα τελευταία αποτελούν απειροελάχιστο τμήμα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα επιπροσθέτως. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης δεν δημιουργούν κανένα είδους βεβαιότητα σχετικά με το πώς ακριβώς πρέπει να υπολογίζουμε τις εκπομπές και όχι μόνο του μεθανίου. Ο εισηγητής θα προτιμούσε λοιπόν να μην επιβληθεί από την αρχή οποιαδήποτε τιμωρία σε αυτή την ε, μικρή κατηγορία οχημάτων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η επανεξέταση που θεσπίζεται με το άρθρο 14 παράγραφος 3 η εναλλακτικά μια αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων μπορεί να διασφαλίσει ότι αμέσως μόλις με, ε, υπάρξει πρόβλημα με την εκπομπή μεθανίου η Επιτροπή θα, θα είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει νέα νομοθεσία. Ε, το ότι δίνει τη δυνατότητα κατόπιν ετοίματο του κατασκευαστή και σε άλλα οχήματα να συμπεριληφθούν στου κανόνε περί ελαφρών εκπομπών αποτελεί θετική πρόθεση τη Επιτροπή. Ο εισηγητή ήταν πρόθυμο να επεκτείνει ακόμα και στι 7, 7 τόνου. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευθούν διπλέ διαδικασίε έγκριση και άλλε περιττέ διοικητικέ ενέργειε. Η αμμονία NH3 εκπέμπεται από βαρέα οχήματα με διζελομηχανές, τα οποία τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εφαρμογής τεχνολογιών επεξεργασίας, που χρησιμοποιούν την ουρδία ως αντιδραστήριο για τη μείωση των οξυδίων του αζότου του Σε περίπτωση βαρέων οχημάτων που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, η αμμονία εκπέμπεται ως φυσικό αποτέλεσμα της κάψη του ίδιου του φυσικού αερίου και όχι για την εξαιρετέρωση των οξυδίων του αζότου, επειδή δεν παράγονται καθόλου τέτοια οξύδια. Η διατήρηση των, ε, του ορίου αμμονίας για βαρέα οχήματα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα θα αποτελούσε την εγκατάσταση ακριβών, ακριβών συστημάτων μείωσης των εκπομπών και αυτό θα αποτελούσε διάκριση σε βάρος αυτής της κατηγορίας ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα, διότι δεν θα επέτρεπε σε εναλλακτικέ τεχνολογίε καυσίμου όπω υγρό, ε, υγραέριο ή φυσικό αέριο να γίνουν οικονομικά βιώσιμε. Η εφαρμογή οριακή τιμή για την αμμονία σε κινητήρε λοιπόν με ηλεκτρικό σπινθήρα για επιβαλλόμενη ανάφλεξη θα πρέπει να αποσυρθεί όπω προτείνει η Επιτροπή. Το εφιστάμενο όριο 10 ppm για οχήματα που ε, απαιτούν ανάφλεξη με συμπίεση ε, αυτανάφλεξη ε, ε, και που αποτελούν την πλειονότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν παραμένει σε ισχύ. Όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. η πρόταση επιδιώκει την προσαρμογή παλαιών διαδικασιών επιτροπολογία στο καθεστώ των κατεξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων όπω ορίζουν τα άρθρα 290 και 91 τη συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τέτοιε πράξει σε σχέση με ευρύ φάσμα κανόνων, διαδικασιών και ορίων που άπτονται τις εφαρμογές των προτύπων Euro 5 και Euro 6. Όπως συμβαίνει με τη μεγάλη πλειοψηφία των πράξεων, η εξουσία έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύων στις 30 Ιουνίου 2019, η οποία αντιστοιχεί στο τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, σε αντίθεση με το προτινόμενο όριστο χρονικό διάστημα. Ε, ισχύουν επίσης οι συνήθεις διατάξεις στην έκθεση της Επιτροπής περί εξουσιοδότηση και περί σιωπηρής παράτασης. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις ε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή απευθεία με τον κύριο Ντες. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. The group, the Κυρία Νταλή η σκιώδης από το νόμο Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατάρχα θα ήθελα να πω ότι στηρίζω έντονα ε, τη λήψη οποιοδήποτε συγκεκριμένου μέτρου βοηθά στη μείωση των ρήπων και βελτιώνει την ποιότητα. Αυτό προσπαθούμε τελικά να πετύχουμε και εδώ. Βέβαια, στηρίζουμε όπως είναι προφανές ε, και τη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να οριστούν αποδεκτά ε, επιτρεπτά όρια για ε, τα αέρια των νέων οχημάτων και την ευθύγραμμιση της νομοθεσίας Ένωσης με νέες τεχνολογικές εξέλιξεις. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι αμφιβάλλω τα μάλλον σε τεφά τις μεθόδους που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είναι η υπερβολική χρήση ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων και την πλήρη απουσία μελετών ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου για πολύ τεχνικά και πολύπλοκα ζητήματα της πρότασης. Ε, υπάρχει επίσης και ανεπαρκής τεχνική αιτιολόγηση στις μελέτες αυτές αντικτύπου για διάφορα ζητήματα. αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε έξι βασικά θέματα. Ξεκινώ με το ανώτατο όριο μάζα. Συμφωνώ με την Κομισιόν που λέει εδώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο, ε, ο ίδιος τύπος ε, οχήματος απαιτεί διπλό έλεγχο, διπλή δοκιμή με τη σημερινή πρακτική. Αυτό συνιστά μεγάλο κόστος και για τον κατασκευαστή ενώ δεν φέρνει και κανένα περιβαλλοντικό όφελος. Ε, προτείνει όμως ο εισηγητής να αυξηθεί αυτή ε, η ανώτατη μάζα στα 7.000 ε, ε, χιλιόγραμμα. Εγώ πραγματικά έχω μεγάλες αμφιβολίες και θα προτιμούσα να παραμείνει η αρχική μάση πρόταση που λέει ότι δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόγραμμα. Και σε ό,τι αφορά τη μάζα του οχήματο, συμφωνώ με την πρόταση τη Κομισιόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα όρια κομπών αμμονίας, έχουμε την πρόταση που λέει ότι πρέπει να εξαιρεθούν ε, τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο. Εγώ θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να διορθωθεί ένα μέτρο που συνιστά διακριτική μεταχείριση ε, κατά των οχημάτων που κινούνται με συμπισμένο φυσικό αέριο και έχει συζητηθεί και ο κανονισμός 595 ε, του 2009 έμεινε εκτός της τελικής έκδοξης του κανονισμού για ανεξήγητους λόγους αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι τα χαμηλότερα ε, εκπομπών ε, θερμοκρασία συγκεκριμένα. Έχουμε για τους ε, υδρογονάνθρακες και το μονοξίδιο του άνθρακα κάποιες τιμές, αλλά δεν είχαμε πρώτα τελευταία χρόνια. Και δεν έχουμε και κάποια όρια σε χαμηλές θερμοκρασίες για τα οξύδια του αζότου. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, συναπόφαση σε αυτό το τομέα. Και σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των οριακών τιμών, αυτό πρέπει να γίνει αφού όμως έχει γίνει για το μονοξίδιο ε, του... Ε, άνθρακα και άλλες ουσίες, κάποια μελέτη. Τώρα, τα όρια για το Euro 6, για τα ελαφρά οχήματα, σε ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου, αυτά είναι, ένα προβληματικ, μια προβληματική, είναι προβληματικές ουσίες μάλλον, γιατί επηρεάζουν την υγεία, ε, ιδίως ε, στα κέντρα ε, των πόλεων. Θέλουμε να έχουμε σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει έμεσα να αυξηθούν οι εκπομπές οξυδίων του αζότου. ιδίως εφόσον έχουμε ήδη κάποιες τιμές που προβλέπονται στον κανονισμό Euro. Εκεί ορίζεται μια οριακή τιμή για τις εκπομπές στο κανονισμό Γιουρσίξ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Επίσης, στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία. Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι μη σημαντικά τα στοιχεία του κανονισμού αυτά που αφορούν τις ωραίες τιμές των εκπομπών. Αυτά πάντοτε αποφασίζονται με συναπόφαση. Τώρα, για την ανάγκη διεξαγωγή μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου για να δούμε το κόστο και το όφελο των ορίων για τα οξύδια του αζώτου είναι σωστό. Πέμπτο, μεθάνιο. Το μεθάνιο θεωρείται θερμοκηπιακό αέριο και πρέπει να θεωρηθεί στο δύναμο διοξιδίου του άνθρωπου. Προβλέπονται ε, οριακές τιμές για το μεθάνο και το γενικά στους συνολικούς ε, υδρογονάνθρακες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προβούμε σε κάποια απορρίθμιση για να μπορεί ε, να ενισχυθεί και η εισαγωγή στην αγορά των ε, οχημάτων με φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, κάποιους κάποια συστήματα ένδειξη και κάποιους μετρητές για το φυσικό αέριο, για τα κύβατα ταχυτήτων. Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσει για την ε, προσαρμογή μετρητών κατανάλωσης καυσίμου, αλλά με την οικολογική οδήγηση νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ε, πρόοδο. Και καλό θα ήταν να έχουμε τα δύο συστήματα μέτρησης ε, και κατανάλωση καυσίμου και για το φυσικό αέριο να τα έχουμε στο όχημα. Υπάρχει τεχνολογία και μπορεί να διατεθεί με μικρό κόστος για το κατασκευαστή σε όλα τα οχήματα και τέλος. Ζητά την εξοδότηση να εγκρίνει τουλάχιστον 10 κατεξότητες πράξεις η Κομισιόν δυνάμει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης. Μειώνει όμως το πρακτικό περιεχόμενο της νομοθετικής πράξης της ίδιας του κανονισμού δηλαδή. Εγώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε αυστήρα στις κανονικές νομοθετικές διαδικασίες. Δεν ε, φαντάζομαι ότι διαφωνεί ο συγγετής και άλλοι σκιώδες θα συνεργαστώ σίγουρα στενά με τον κύριο Ντές. Thank Θα σε ευχαριστώ πολύ κύριε Ανταλή. αλλά να παρακάσω τους υπόλοιπους ομιλητές να μιλάνε πιο αργά για να διευκολύνεται η μετάφραση. Θα προσπαθήσω να μιλήσω εγώ πιο αργά. Λέω ο κύριο Γερμπράντη. Ο Νίλ Στόρβαλτ που ήταν ο συζητητής δεν μπορεί να παραστεί. Μου ζήτησε λοιπόν να τον εκπροσωπήσω σήμερα. Έχω λοιπόν κάποιε παρατηρήσει. Πρώτον, ο βασικό στόχο είναι οι εκπομπέ οξυδίων του αζότου. Και είναι ένα πολύ καλό στόχο σίγουρα η μείωση αυτών των εκπομπών. Αν δείτε ιδίω την έκθεση τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία τη προηγούμενη εβδομάδα, που δίνεται έμφαση για μια ακόμη φορά στο τεράστιο κόστο που έχει για την κοινωνία η ατμοσφαιρική ρήπανση. Υπολόγισαν με βάση πολλά δεδομένα το συνολικό κόστο τη ατμοσφαιρικής ρήπανση στην Ευρώπη σε 1,4 τρισεκατομμύρια ε, ευρώ. Και στην αιτιολογική έκθεση του εισηγητή, παρόλα αυτά, εκπλήσωμε γιατί λέει ότι καταρχήν χαιρετίζει μέτρα για τη βελτίωση ε, της ε, ποιότητας του αέρα. Αλλά κάνει κάποιες προτάσεις, τι να πω, ε, είναι σημαντικό το θέμα και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών και αλλού όπου συζητούμε την ποιότητα του αέρα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Με εκπλήσει επίσης η παρατήρηση πάντα στην ετολική έκθεση ε, σε σχέση με την αυτοκίνητο βιομηχανία. Παραλαμβάνει τη ιστορία από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ακούμε πάντα ε, κινδυνολογίες ε, όταν μιλάμε για τα ε, κατώτατα, κατώτερα όρια εκπομπών από την αυτοκινητοβιομηχανία. λέει δεν πρόκειται ποτέ να τα πετύχει ε, και πάντα βλέπουμε ότι με το παραπάνω είναι ικανοί να τα πετύχουν. Αν δείτε τις εκπομπές του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, το 2014 ήδη οι στόχοι έχουν υπερβεί, τις έχουν υπερβεί οι βιομηχανίες ήδη και από, πιο καλά είναι τα, ε, οι επιδόσεις τους από αυτές που προβλέπονται για το 2015. Σε αυτή την έκθεση τώρα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ισορροπία πράγματι. Αυτό είναι και το μήνυμα του κ. Τόρβαλ του σκιώδου εισηγητή μας. Εκ μέρους της Άλντε θα καταθέσουμε ορισμένε τροπολογίες. Προσβλέπουμε όμως μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ, σκιώδης από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν τον τεράστιο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και υπάρχει και η πρόσφατη μελέτη που αναφέρατε που έγινε από τον ΠΟΗ που, λέει, θέτει το θέμα του οικονομικού κόστους της ρήπανσης και το ανεβάζει στο 1,63 το χρόνο. Αυτό το κόστος παίρνει τη μορφή 600.000 πρόωρων θανάτων κάθε χρόνο και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων νοσούν από την ρήπανση των αυτοκινήτων που προκαλούν τα αυτοκίνητα. Ε, πολλοί έχουν σύγχυση στο μυαλό τους σε σχέση με τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα που έχει κέρια σημασία αλλά έχουν σύγχυση και σε σχέση με το γεγονός ότι τα αέρια που βλάπτουν το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα προέρχονται από τις μεταφορές κυρίως. Αν μειωθούν αυτοί, αυτές οι πηγές μόλυνσης, αυτό ε, είναι σημαντικό. Στα πλαίσια των προτύπων Euro 5 και 6 που προσφέρουν μια ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό. Ε, θέλουμε παγκόσμια αποτελέσματα. Η πρόταση της Κομισιόν δεν αναφέρει όμως ε, κανένα μέτρο που θα εμείωνε ουσιαστικά τις εκπομπές, αναφέρεται σε μέτρα ευελιξίας για τους κατασκευαστές στα κράτη-μέλη. Διάφορα θέματα σημαντικά όπως η ε, εξαιρέσεις για τα οχήματα αερίου και η ουσιοδότηση πράξη που προτείνεται. Ε, δίδεται προτεραιότητα στα τελευταία αφαιρώντας ε, τα όρια εκπομπών αμμονίας, ε, βάζοντας για το μεθάνιο ε, ισοδύναμα του ε, διοξιδίου του άνθρακα, ε, προσαρμόζοντας τις, τους συνολικές εκπομπές υδρογονανθράκων. Ε, όμως ε, όλα αυτά επηρεάζουν ε, περισσότερο και από το διοξίδιο του άνθρακα. υπάρχει διαρροή μεθανίου που είναι σημαντικό αέριο θερμοκηπίου. Σίγουρα θα πρέπει να ε, έχουμε μια ε, προσέγγιση ουδέτερη ως προς την τεχνολογία. Η Κομισιόν προτείνει να τεθούν διάφορα όρια εκπομπών με κατεξουσιοδότηση πράξης. Όμως ε, δεν κάνουν παράλληλα εκτιμήσεις επιπτώσεων. Αυτό είναι ανεπαρκές και δεν μας ενημερώνει αρκετά ούτως ώστε να εξουσιοδοτήσουμε σχετικά την Κομισιόν. Αυτές οι προτάσεις έχουν πολύ χαμηλούς στόχους και ως Επιτροπή ε, ε, Περιβάλλοντος δεν ε, μπορούμε εύκολα να συμφωνήσουμε μέχρι που θα έλεγα να απορρίψουμε την έκθεση. Και ο εισηγητής δεν βελτιώνει την κακή ε, πρόταση της Κομισιόν για να μειώσει τις επιβλαβείς εκπομπές. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, σχετικά με υποχρεωτικούς δείκτες και μετρητές κατανάλωσης καψίμων για κάποιες κατηγορίες οχημάτων. Γιατί έτσι θα ενθαρρύνονται οι οδηγοί να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων με, λίγο με μικρό επενδυτικό κόστος ε, υποχρεωτικοί δείκτες και οι μετρητές κατανάλωσης καυσίμων μπορεί να ε, βελτίωναν την ε, μελέτη επιπτώσεων, όμως δεν εμφανίζονται στην πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι στις διαδικασίες δοκιμών για τις εκπομπές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις. Συλλέγει μια δράση να μην, να μην υπάρχουν κάποια μέτρα αποθετικά για να μην χρησιμοποιείται το μεθάνιο σαν καύσιμο. Τα ορυκτά καύσιμα, ε, όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει ελάχιστο άνθρακα και τα οχήματα με μεθάνιο ε, συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του δεξιού του άνθρακος και των σωματιδίων από τους ρηπαντές τους, ε, πιο, τους λιγότερους που δεν φαίνονται τόσο πολύ. Για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να μειώσουμε και την εκπομπή του μεθανίου. 70 φορές μεγαλύτερο ε, αποτέλεσμα έχει από τον άνθρακα σε μια μεγάλη χρονική περίοδο προτείνεται να αυξηθεί και η μάζα των αυτοκινήτων που καλύπτονται από το, διά, από το μέτρο αυτό στους 7,2 τόνους. Ε, εκτιμούμε και την πρόταση του συγητού να καθοριστεί πιο συγκεκριμένο όριο όσον αφορά την εξουσία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κατεξοδότηση πράξης. Πιστεύουμε όμως ότι είναι ένα από τα νομοθετικά κείμενα για τα οποία η κατεξοδότηση πράξη θα τροποποιήσουν ε, ουσιαστικά τμήματα του τροποποιημένου κανονισμού. Ένα στοιχείο που μας κάνει θεωρούμε να μην δίδεται τόση εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα μπορεί να εντοπίζει νέα όρια μέσω της ε, κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Πρόκειται περί προτάσεως ε, που θα εντοπίζει τα όρια των εκπομπών το οποίο δεν είναι δευτερεύουσης σημασίας στοιχείο και δεν θα ήταν σκόπιμο να το αφήνουμε, να το αφήνουμε στη, τον καθορισμό αυτών των ορίων στις πράξη. Σε ευχαριστώ. Και τώρα τα μέλη της Επιτροπής θα πάρουν το λόγο. Μόνο ένα θέλει το λόγο. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ζήτησα τον λόγο γιατί είναι τεχνικός ο φάκελος, αλλά εγώ είμαι και στην Επιτροπή Μεταφορών και το χειρίζομαι το θέμα για την ομάδα μου. Κάποια σχόλια, πολλά είπαμε ήδη, πράγματι είναι πολύ σωστό η ε, ποιότητα της ατμόσφαιρας ε, όντως ε, επιβαρύνεται από τα οχήματα και στην ναυτιλία ασχολήθηκαν με τα οξύδια του αζότου και προέβησαν σε μέτρα. Τώρα το μεθάνιο, όπως είπε και ο συνάδελφος Τέιλορ, από μόνο του δεν είναι βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, αλλά επηρεάζει και αυτό το κλίμα και πολύ αποφασιστικά μάλιστα. Ε, πάντως στην περίπτωση αυτή, την πρόταση του κυρίου Ντες, γιατί το μεθάνιο εκπέμπεται εδώ από χήματα που χρησιμοποιούν αέριο, πράγματι το μεθάνιο είναι πολύ μικρό ποσοστό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη κατασκευή, να υπάρχει και μια υποδομή για εναλλακτική και εναλλακτικά κάψιμα και υγραέριο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα οχήματα που θα τα χρησιμοποιούν και εκεί θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την εκπομπή μεθανίου αλλά ακόμα είναι πολύ μικρός ο τομέας αυτός ο, τα, ο αριθμός αυτών των οχημάτων τρίτον για την οικολογική οδήγηση, eco-driving, βεβαίως είναι πολύ λογική και καλή πρόταση που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ε, και να διδάσκεται και στις σχολές οδήγησης. Είναι καλή προσέγγιση, ε, τεχνικά μπορεί να γίνει και όλοι οι οδηγοί θα καταλαβαίνουν καλύτερα πώς μπορούν να οδηγούν σωστά χωρίς να επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Πολύ σωστή η πρόταση λοιπόν αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Οπότε Α, να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πετινέλη, αν έχει την καλοσύνη, ας εκφράσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Προέδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να συμμετάσχω στην παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως ε, του εισηγητού του κ. Ρης και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προετοιμασία του σχεδίου εκθέσεως που κατά την άποψή μας σε μεγάλο βαθμό μοιράζεται τις προθέσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπής να αντιμετωπιστούν οι τομεί εκείνη των, ελαφρών, των νομοθεσία για ελαφρέ και πιο, βαρι... πιο σημαντικές εκπομπές για να εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον. Τώρα ακροθυγώς να σχολιάσω κάποιες τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο εκθέσεως. Καλωσορίζουμε τη στήριξη του συγκητού για την αύξηση της για την ε, έγκριση οχημάτων λόγω αυτών των μέτρων χωρίς μείωση του επίπεδου περιβαλλοντικής προστασίας και να μην δημιουργούμε άχθος για την... μειώνουμε το άχθος για την αυτοκινητοβιομηχανία. Όσον αφορά τις κατεξουσοδότησης εν πράξεις, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταχική πρόταση είναι πλέον δεδειγμένη για τις εξουσίες που τις χορηγούνται. Κατανοούμε όμως την πρόθεση ηγητού να περιοριστεί η περίοδος και να δοθεί παράταση βάση της εκθέσεώς μας. Η πιο προβληματική τροπολογία για μας είναι η άρση της μεθοδολογίας για υπολογισμό του αντιχτύπου των νερίου του θερμοκηπίου και κυρίως του μεθανίου σε ισοδυναμία με διοξείδιο του άνθρακος. Λαμβάνουμε υπόψη την τροπολογία, θεωρούμε όμως ότι η πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου ε, δεν είναι πλήρως κατανοητή και δεν καλύπτει τα πάντα. Η αρχή της ισοδυναμίας διοξιδίου του άνθρακος εισήχθη για να λάβουμε υπόψη τα αέρια του θερμοκηπίου όσον αφορά το μεθάνιο και να μειωθούν εκπομπός του μεθανίου όταν έχει αυξηθεί το συνοδικό όριο των υδρογοναθράκων. Θέλουμε να αξιολογήσουμε τις περαιτέρω συνέπειες που μπορεί να έχει προτάσει το Ευρωκοινοβουλίο. Κατανάλωση καυσίμων και δείκτες για την αλλαγή ταχυτήτων αυτοί οι μηχανισμοί μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων περισσότερο, παρά τις εκπομπές. Ίσως καλύτερη θέση θα είχαν τα μέτρα στον κανονισμό για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διοξιδίου του άνθρακος, παρά εδώ. Εδώ ο στόχος αφορά τους ρηπαντέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετινέλη. Ο κύριος Λίντς έχει ξανά το λόγο. Πολύ σύντομα να συνοψίσω βέβαια δεν θέλω να προδικάσω αυτά που θα πει ο εισηγητής ε, ως προς την ουσία ε, πάντως βλέπω ότι χρειάζεται ακόμα κάποια συζήτηση για το μεθάνιο για παράδειγμα Βλέπω όμως να συμφωνούν για την εξουσιοδότηση πράξη, για, τη, για και το, το νάζ των οχημάτων που πρέπει να συμμετέχουν στη ρύθμιση. Ε, είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής ε, μετά από την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών θα συζητήσει μαζί σας και σίγουρα θα βρεθεί και λύση συμβιβαστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίντς. Τώρα, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 19η Μαΐου, το μεσημέρι στις 12. Η εξέταση των τροπολογιών, αν υπάρξουν, είναι 25η Ιουνίου. Η έγκριση στην Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι η 15η Ιουλίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια αναμένεται στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου 2015. Προχωρούμε και πάμε στο επόμενο σημείο, το οποίο αφορά την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αυτό είναι στενά συνδεδεμένο θέμα με το προηγούμενο. Καταρχήν να δώσω το λόγο, το λόγο στην συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα επόμενα 40 χρόνια πάνω από 2,5 δις άνθρωποι θα κατοικούν σε πόλεις. Το 90% του πληθυσμού θα είναι σε αναδυόμενες σε, στις πόλεις των αναδειωμένων οικονομιών, αναπτυσσομένων χωρών, έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα προς επίλυση όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική, όσον αφορά την αστικοποίηση και την κινητικότητα που συνδέεται με αυτό. Στην Ευρώπη το 70% του πληθυσμού ζήτησης της πόλης και συνέπειε των δημογραφικών μεταβολών κοινωνικονομικών αλλαγών όπως η γύρανση του πληθυσμού η μετανάστευση σαφώς ε, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και θα καθορίσουν καταστάσεις και περιστάσεις διαφορετικές. Βάση των προσεγγίσεων, 90% των Ευρωπαίων κατοίκων εκτίθεται σε συγκεντρώσεις πάνω από το ασφαλή όσον αφορά τη ρήπανση. Είναι ένα στοιχείο που μας κάνει να προβληματιζόμαστε και διαφαίνεται το γεγονό ότι το 96% των μεταφορών στην Ευρώπη εξαρτάται ακόμα από το πετρέλαιο και τα παραπροϊόντα αυτού. Παράδοξο είναι αυτό. 45% των κατοίκων μετακινείται εντός των πόλεων σε αποστάσεις λιγότερες από, το, 5 χιλιόμετρα και 40% κάτω από 20 χιλιόμετρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι πόλεις πρέπει να δώσουν μια απάντηση στο πρόβλημα της κινητικότητας. Και στις πόλεις το πρόβλημα της συμφόρησης μεταφράζεται με διαφορετικές συνέπειες αρνητικές για το περιβάλλον και για την πόλη. Ε, η μόνη ατμόσφαιρα καταρχάς, το συζητήσαμε πριν, στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, 23% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο είναι στατικέ εκπομπέ και από τον τομέα των μεταφορών. Αλλά και η χορύπανση από τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντο βλέπουμε ότι σπάσαμε ρεκόρ. Ότι αντίκτυπο στην υγεία όσον αφορά την χορύπανση είναι οφείλεται στο 90% των υποθέσεων που συνδέονται μάλιστα τα προβλήματα με την χορύπανση από την ε, κυκλοφορία των μεταφορών είναι και θέμα ασφάλειας. Ε, στην Ευρώπη ε, είχαμε λευκή βίβλο για την ασφάλεια των μεταφορών, έχουμε ψηφίσει διάφορα ψηφίσματα, έχουμε και το Urban Mobility Package που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ενώσης. Η εφαρμογή όμως των στρατηγικών απαιτείται από τα κράτη-μέλη και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αδεφισβήτητο ότι το ΙΟΤΑΧΗ είναι το βασικό μέσο μεταφοράς, το πιο διαδεδομένο, το πλέον χρησιμοποιούμε κατά μέσο όρο 50% στην Ιταλία. Δυστυχώς είμαστε 69% της χρήσης του ΙΟΤΑΧΗ σε σχέση με άλλα μεταφορικά μέσα. 16% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα μεταφοράς και μόνο το 12% το ποδήλατο. στην γνωμοδότηση που ετοιμάσαμε, στο κείμενο, θεωρήσαμε σημαντικό να τονίσουμε την τηλεργασία. Τη δυνατότητα δηλαδή να μειωθούν οι φυσικές μετακινήσεις εντός των πόλων, προωθώντας πολιτικές που αφορούν την τηλεργασία ηλεκτρονική εκμάθηση, e-learning, διάφορες λύσεις που μας προσφέρει η τεχνολογία. Eh, ehm, λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής των σωστών υποδομών, δημιουργίας των σωστών υποδομών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ένα τα παραδείγματα τα συγκεκριμένα με θετικά αποτελέσματα πρέπει να προωθούνται. Τα δίκτυα δημοσίου φωτισμού αν χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να έχουμε διαδεδομένη υποδομή για να προωθήσουμε την χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και να εγκαταλείψουμε τα οχήματα με ορυκτά καύσιμα. Σίγουρα είναι ουσιαστικό να δυσκολίσουμε τα συστήματα τα διατροπικά των μεταφορών, να υπάρχουν ζώνες που είναι διαθέσιμες στα μαζικά μέσα μεταφοράς και στα ηλεκτρικά και να υπάρχει car sharing και τα ποδήλατα, χρήση ποδηλάτων, η σωστή προσέγγιση για να αλλάξουμε τον τρόπο κινητικότητας της πόλης. Όχι μόνο αυτό, προτείνουμε και τροπολογία τροποποίηση τη αλλαγή τη Σύμβαση τη Βιέννη για την οδική κυκλοφορία ούτως ώστε να προηγούνται των άλλων μέσων μεταφοράς τα ποδήλατα στην κυκλοφορία και έτσι μπορούμε να αλλάξουμε ένα από τα παραδείγματα αλλαγή του τρόπου κινητικότητας και αναθεώρηση του οδικού κώδικα, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να προστατεύουμε καλύτερα τους αδύναμους. Και να προωθήσουμε την κινητικότητα τη σωστή. και τι γίνεται με την προκήρυξη διαγωνισμών για τι υπηρεσίε μεταφορών και την όλη οργάνωση των μεταφορών, να υπάρχουν κριτήρια βιωσιμότητα που επικρατούν εκεί. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για λύσεις που δίνουν τη η αξία στον αφορά το περιβάλλον και την κοινωνία. Αν δεν γίνει αυτό, η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει που θα είναι δυσάρεστη. Αυτές είναι βασικά οι προτάσεις που προβάλλουμε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η ριζική αλλαγή της νοοτροπίας για την κινητικότητα περνά και από αλλαγή του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών. Είναι σαφές ότι η συμπεριφορά των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Η επιλογή που κάνει ο κάθε πολίτης. Πρέπει να αλλάξει ριζικά. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται κίνητρα για τον πολίτη. Πρέπει να ζήσει την αλλαγή σαν κάτι θετικό. Έχουμε δύο μοχλούς, την ευαισθητοποίηση πρώτα απ' όλα, Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα, δεν πάει συνεχιστεί αυτό. Και μετά ένα μοχλό που χρησιμοποιηθεί είναι οικονομικό. Δηλαδή το πόσο είναι βολικές οι δημόσιε συγκοινωνίε, που θα μπορούσαν να είναι και δωρεάν. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο. Μη λησμονούμε και τη συμμετοχική διαχείριση κινητικότητας. Οι πολίτες των πόλεων είναι εκείνοι προς οποίους πρέπει να απευθυνθούμε. Να μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση κινητικότητας. Αυτό μπορεί να είναι κάτι θετικό για τις πόλεις. Να δίδονται κίνητρα μέσω των συστημάτων που θα χρησιμοποιούμε που θα βραβεύουν τις σωστές α, συμπεριφορές. Με τα χαρά διαπιστώνω ότι οι εθνικές πολιτικές που στηρίζουν βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις μπορούν να ωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία μόνο κατόπιν υποβολή συγκεκριμένου σχεδίου. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Η χρηματοδότηση και η χρήση των ταμείων συνοχής και των εθνικών ταμείων απαιτούν και την υποβολή βιωσίμων σχεδίων. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και είμαι σίγουρη ότι τελικά μπορούμε να κάνουμε έξοχη δουλειά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Εύη. Σκιώδης από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. και Μπριάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαντλητική της έκθεση. Συμμερίζομαι την ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί. Έχουμε μία έκθεση με πολλές θετικές πτυχές. Πρέπει να εκφράσουμε τη θέση Επιτροπής Περιβάλλοντος, να επικεντρωθούμε επί των θεμάτων που άπτονται του περιβαλλοντικού. Ο περισσότερος πληθυσμός στην Ευρώπη βρίσκεται σε μεγάλες πόλεις, εκεί ζει, οι μεταφορές των ατόμων είναι σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας, είναι κάτι θετικό, μας επιτρέπει να φτάσουμε στις εργασίες, να έχουμε παροχή σε υπηρεσίες, ε, δραστηριότητες ε, ε, καλλιτεχνικές, τουριστικές κλπ. Αυτή η κινητικότητα και οι μεταφορές, κυρίως οι αστικές, θα πρέπει να γίνουν όλο και πιο βιώσιμες από πλευρά κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές στοιχές, η κινητικότητα έχει πολλές σχέσεις με τα περιοδικά στοιχεία που συζητούμε, διότι το μέσο των μεταφορών είναι υπεύθυνο για περίπου το 1 τρίτο της κατανάλωσης ενέργειας και αυτό είναι στοιχείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και πάνω από το 1 πέμπτο των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, των αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε από αυτού. Οι μεταφορές είναι και όπως υπόθηκε πηγή και άλλης ρήπανσης ατμοσφαιρικής όπως σωματίδια και η Δεν παραγούν μόνο τα μέσα μεταφοράς στη ρήπανση, αλλά και τα οχήματα, τα άλλα, τα γιοταχή. Πολλά άτομα δυστυχώς, λόγω ατομικής συμπεριφοράς, προτιμούν το γιοταχή σε σχέση με τις δημόσιες κοινωνίες και τα γιοταχή στις πόλεις κατέχουν και χώρο και δημιουργούν και επιδείνωση τεστικού περιβάλλοντος ε, και εμποδίζουν και τους πεζούς γιατί καταλαμβάνουν χώρο. Χρειάζονται οδικές υποδομές να δημιουργηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τον αντίκτυπο για το περιβάλλον γιατί καταναλώνεται έδαφος. Βγήκε μια έκθεση της Ίσπρα για την Ιταλία όσον αφορά την κατανάλωση εδαφών. Είναι θεμελιώδε ζήτημα, δυστυχώς είναι πάντα πολύ μεγάλη αυτή η χρήση των εδαφών και έχει και μεγάλη επίδραση στην ύπεθρο και στο τοπίο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μέσω τροπολογιών ε, θα το ανακαλύψουμε. Ε, συμφωνούμε πολλά από αυτά που αναφέρει η συγκήτρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθούν ε, το περπάτημα, το ποδήλατο κλπ. Να, να αλλάξει ο τρόπος ζωής, να μειωθεί η κυκλοφορία κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που πρέπει να δρομολογηθούν και μπορούν. Και τελικά καμή, τίποτα από τα μέτρα δεν, αυτά δεν είναι κάτι ε, εξαντλητικό αλλά και χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου μετακίνησης της πόλης και μια ληστική προσέγγιση και αλλαγή νοτοπίας. από πλευράς ΕΛΚ η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Δεν μιλώ εκ μέρου ε, σε καμία περίπτωση του ουσιώδου του ΕΛΚΑ. Να πω όμω ότι άκουσα με πολύ προσοχή την εισηγήτρια και θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα την παρέμβασή της, γιατί ήταν πάρα πολύ διεξοδική. Αυτό το ζήτημα της, αστικής, ε, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει εδώ και καιρό γιατί και 25 χρόνια εκλεγόμουν σε σύμβουλο σε μια πόλη μεγάλη και είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται κάθε τρεις και λίγο. Γιατί το ζήτημα των μεταφορών έχει να κάνει και με τη ρήπανση των μεγαλού πόλεων και περνάει ε, σίγουρα ε, από την αύξηση των ε, συγκοινωνιών γιατί είναι τόσο μεγάλο το κόστος της κατοικίας στο κέντρο της πόλης που όλο και περισσότεροι συμπολίτε μας ζουν στην περιφέρεια. Άρα μας δημιουργεί αυτό μεγάλο πρόβλημα συγκοινωνιακό πρέπει να λύσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά βιώσιμη κινητικότητα πρέπει σίγουρα να αναπτύξουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πολύ περισσότερο που θα πρέπει να είναι και καθαρές αλλά και αποτελεσματικές ασφαλής επίσης, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και θέματα ασφάλειας ε, σε κάποιες ώρες της ημέρας ή της νύχτας. Άρα εμείς πρέπει να τα δούμε αυτά τα προβλήματα. Εμείς είμαστε στην Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος, άρα μας απασχολούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα της ποιότητας του αέρα, της ατμοσφαιρικής πίεσης και τα προβλήματα υγείας. Άκουσα ότι υπάρχουν καλές πρακτικές που θα πρέπει να προταθούν, μάλιστα. Αυτό θα είναι πολύ καλό και για την υγεία Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε απόλυτα τις προτάσεις της εισηγήτριας και να συμφωνήσουμε με την ανάλυση της. Τα κίνητρα ανάπτυξη υποδομών είναι και αυτό σημαντικό, η χρηματοοικονομική υποστήριξη. Τουλάχιστον στη χώρα μου σήμερα ξέρουμε ότι ε, οι πόλεις, τα αστικά κέντρα πρέπει να αναλάβουν όλο και περισσότερα πράγματα, άρα έχουν όλο και περισσότερες οικονομικές δυσκολίες, άρα χρειάζεται η στήριξη της Ευρώπης, που ήδη παρεμβαίνει εδώ και καιρό, το έχω δει και στη δική μου την πόλη, με την ανάπτυξη του τραμ, για παράδειγμα, που το υποστήριξε η Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε τελικά να φτάσουμε σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τη συγκοινωνία στα αστικά κέντρα. Νομίζω ότι θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις της εισηγήτριας και νομίζω θα τις στηρίξουμε στο μεγαλύτερό τους μέρος. Θα δούμε βέβαια κατά πόσον θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και εμείς κάποιες λεπτομέρειες, κάποια μικροπράγματα από πλευρά ΣΕΛ. ευχαριστώ πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ από την Άλντε. Κυρία Μάστερ, επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια, συντάκτρια. Η αστική βιωσιμότητα είναι θέμα της Επιτροπής Μεταφορών, όπου είμαι. Και μπορεί κανείς να κάνει στην αστική βιωσιμότητα πολύ περισσότερα πράγματα και να λάβει πολύ περισσότερο υπόψη το περιβάλλον από ό,τι γενικότερα. Γιατί η αστική βιωσιμότητα έχει άλλες δυνατότητες από τη βιωσιμ... η... κινητικότητα στην ύπεθρο. Ε, το ξέρω αυτό εκ Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, σωστή ε, διεύθυνση της κυκλοφορίας. δεν ξέρω και ακριβώς τι εννοεί αυτό γιατί και εδώ υπάρχει ψηφιοποίηση και ήδη μπορούν να γίνουν πολλά για να αποφεύγονται τα μποτιλιαρίσματα. Αυτό βέβαια είναι μια πλευρά του νομίσματος. Το άλλο είναι η ηλεκτρική κινητικότητα, πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε πάντοτε ότι είναι σημαντικό να δούμε και την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι ηλεκτρική ενέργεια, ε, πρέπει να δούμε από πού προέρχεται και εξασφαλίζεται, γιατί αλλιώς ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αηφόρος από μόνη της. Να το δούμε λοιπόν και αυτό, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά, ε, τα οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική για την αστική βιωσιμότητα του μέλλοντος. Πολλές ε, φορές ε, ακούμε για καινοτομίες που θα γίνουν ε, και που μπορεί ενδεχομένως να αυξήσουν τόσο πολύ τον αριθμό των ποδηλάτων που να ε, ε, εξαντληθούν οι δυνατότητες. Υπάρχουν όμως και οι δυνατότητες να αποθήκευσης και φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων πολλές φορές δωρεάν και για τα αυτοκίνητα και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Θα πάρει χρόνο για να εφαρμοστεί αυτό, αλλά είναι πολύ καλό παράδειγμα παρόλα αυτά και αυτό είναι βιώσιμο 100%. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε, ε, είναι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν κάπου και πρέπει να ε, γίνουν ευρύτερα γνωστές. Ε, επίσης Clean Power ε, ε, for Transport, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε γιατί θα εφαρμόζεται όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Κάτι άλλο πολύ καλό που το λέει η συντάκτρια και είναι καλό για το περιβάλλον, δηλαδή και τις εκπομπές, είναι το car sharing, να μοιράζεται κανείς το αυτοκίνητο και άλλες συμμετοχικές μορφές μεταφορών, πολύ καλό και μπορεί να γίνει και στην πόλη. Είμαι επιφυλακτική λίγο ε, να δώσουμε γενικά προτεραιότητα στα ποδήλατα έναντι των ε, αυτοκινήτων. Πώς ε, μπορεί να γίνει αυτό, είναι πάρα πολλά τα μεταφορικά μέσα, σίγουρα θα πρέπει και μπορεί στις πόλεις να αυξηθεί ο αριθμός των ποδηλάτων που χρησιμοποιούνται, είναι καλό και για την υγεία, όχι μόνο για τα ηλεκτρικά αλλά και τα κανονικά αλλά και για τα δίκυκλα γενικότερα, θα πρέπει όμως να δούμε τι προϋποθέσεις υπάρχουν ανάλογα με την ε, κυκλοφορία στις πόλεις και να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα ποδήλατα. Κάτι άλλο που δεν αφορά τόσο το περιβάλλον αλλά είναι μια πρόκληση, το UPNV που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο γιατί είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένο για τα εισιτήρια και στην Επιτροπή Μεταφορών υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλία για αυτό το σύστημα. Υπάρχουν κάποιε πόλει που έχουν ήδη εξαιρετικά μοντέλα. Ξέρω ότι τα καλύτερα είναι στη Γερμανία, στο Αμβούργο, που δεν χρειάζεται κανεί καθόλου το αυτοκίνητο γιατί οι δημόσιε μεταφορέ, οι κοντινέ αποστάσεις είναι τόσο καλά δομημένες που με ένα εισιτήριο μπορεί να πάει κανεί παντού. Οπότε δεν μπαίνει στον πειρασμό να πάρει το αυτοκίνητό του γιατί πάει πολύ πιο γρήγορα με τα δημόσια μέσα μεταφορά, ε, ακόμα και αν δεν σκέφτεται το περιβάλλον δηλαδή. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό. Ποιε πόλει έχουν ποιε καλέ και θετικέ εμπειρίες και τι μπορούμε να μάθουμε από του άλλου. Και, υπάρχει κάτι και υπάρχουν και καινοτόμα ε, συστήματα όπως ένα ε, ο εναέριος ε, που κινείται με σύρματα και ε, θεωρείται ακόμα λίγο εξωτικό γιατί ε, ε, είναι ένα αέριος όπως λέει και η λέξη, κρέμονται εκεί από πάνω. υπάρχει όμως δυνατότητα να το εξετάσουμε και αυτό είναι καλό να ασχολείται η Επιτροπή Περιβάλλοντος με όλα αυτά που άπτονται μεν των μεταφορών αλλά αφορούν και το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι ε, τα τελευταία, αυτά ε, τα ε, οχήματα, τα εναέρια τα βλέπω λίγο έτσι κάπως με φόβο αλλά τέλος πάντων Προσβλέπουμε στη γνωμοδότηση ε, της εισηγητρίας και την ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά της. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφορών και υγείας, συγκοινωνιών και υγείας, γιατί επηρεάζουν οι συγκοινωνίες την υγεία όλου του πληθυσμού και άμεσα αλλά και με την ρήπανση του περιβαλλοντος χώρου τους, όπως μεταξύ άλλων ε, δημιουργούν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της ατμοσφαιρικής πύρασης, ε, ρήπανσης ε, και η χορύπανση από τα αεροπλάνα ή τα τρένα επίσης ένα θέμα. Στη Βέρνη, στο Πανεπιστήμιο, έγινε μια μελέτη και λέει ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 60 δεσιμπέλ είναι η χωστάθμη λεει οτι κατα μεσο ορο τουλαχιστον 60 συμπέλη ειναι η θορυβου ιδίως για αυτούς που ζουν κοντά σε αεροδρόμια και 30% περισσότερο κινδυνεύουν να πεθάνουν από ε, καρδιακή ανακοπή. Στο Λονδίνο, ε, στο Χίθρο, πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι ε, που είναι κοντά, ζουν κοντά σε αυτούς τους διαδρόμους, πτήσεις, κινδυνεύουν και χρόνια εκτεθειμένα στους κινδύνους αυτούς παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα, ελληματική προσοχή, μνήμη, επίλυση προβλήματος, απάτη τηλεφώνου, όχι λάθος. και η απόκτηση ικανοτήτων ε, ανάγνωσης. Ξέρουμε ότι οι οδικές μεταφορές είναι η βασική πηγή ε, πυρήπανσης, ε, βλάπτει και το περιβάλλον και την υγεία μας και κακή ατμοσφαιρική ο κακός ατμοσφαιρικός αέρας δημιουργεί, έχει προκαλεί και πολλούς πρόωρους θανάτους. Υπάρχει οικονομικός αντίκτυπος που δεν τον έχουμε ε, εκτιμήσει απόλυτα. Πρέπει να τονίσουμε τη σχέση οικονομικού αντικτύπου και υγεία, γιατί υπάρχει και πιστεύω ότι στα αστικά κέντρα έχουμε τις καλύτερες ευκαιρίες και δυνατότητες να κάνουμε τη διαφορά και να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο για τη βιώσιμη χρήση των πόρων και του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το αισθημόμενο ιατρικό κόστος, το υπολογίζει σε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Είναι γύρω στο 1 δέκατο όλου του ΕΠ της Ένωσης. Αυτό το ποσό. Επίσης είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ως προς το τι είδους επιβλαβής ρήπαση προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Τα ε, σωματίδια, παραδείγματο χάρη, η ρήπη, ε, η διοξυδία του άνθρακα που εκπέμπουν οι εξατμίσεις. Και σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί η προσέγγιση πολλών δήμων και πόλεων και κρατών για το ντίζελ για παράδειγμα και τη χρήση της ολοκίνητων οχημάτων στις πόλεις. Η βιωσιμαστική κινητικότητα περιλαμβάνει μέτρα για το πρασίνισμα των πόλεων, τον εφήχορο ταξικό σχεδιασμό, όλα αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και για την υγεία που δημιουργεί η ατμοσφαιρική ρήπανση και η χορύπανση. Επίσης, σχέση μεταξύ κλιματικής πολιτικής και μεταφορών. Πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Αν δεν εστιάσουμε περισσότερο σε εκπομπές αυτές από το τομέα των συγκοινωνών και των μεταφορών, οι συνολικοί στόχοι για το κλίμα δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν γιατί οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας όπου οι εκπομπές αερίου των θερμοκηπίου αυξάνονται συνεχώς κατά 30% τα τελευταία 25 χρόνια. Και μόνο εάν έχουμε πιο ολοκληρωμένες πολιτικές και προσεγγίσεις ε, με αλλαγή τρόπων ε, μεταφορών, με εναλλακτικά καύσιμα, με μείωση του όγκου των μεταφορών. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε, να πετύχουμε αυτό το στόχο. Σίγουρα θα συμμετάσχω και εγώ στην κατάρτιση της έκθεσης και ευχαριστώ πολύ την κυρία Εύη για τη δουλειά της μέχρι τώρα. Thank you very much. And after becoming a... Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πλέον να αντιληφθεί την άποψη των σκιωδών και πηγαίνουμε στους υπόλοιπους ε, ομιλητές ε, και αντογανώ. Καταλαβαίνω και ακούω τις καλές προθέσεις, άκουσα και διάβασα και με προσοχή την ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να επιμείνουμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, πολύ σημαντικότερο από τις διάφορες ιδέες για τις βιώσιμε μεταφορές και συγκοινωνίες. Τι μοντέλο κοινωνίας και κοινωνιοτεχνικής οργάνωσης θέλουμε. Προτείνει η Κομισιόν ρύθμιση της πρόβασης ε, στα αστικά κέντρα, συλλογή πληροφοριών ε, και περαιτέρω εξυγχρονισμό με λύσεις όλο και πιο καινοτόμες όμως για να πετύχουν αυτοί οι μετασχηματισμοί είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα μεταφορών και κινητικότητας ολοκληρωμένο, διασυνδεδεμένο. Και για να ρυθμιστεί ένα τέτοιο σύστημα, τα κράτη-μέλη και ένωση θα πρέπει όλο και πιο πολλούς κανόνες ε, να εκπονούν. Και αυτό βλέπουμε ότι είναι ε, ακόμα ε, μεγαλύτερη γραφειοκρατία ίσως και υπερβολική. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην τοπική, ρεαλιστική αλλαγή επιτόπου και να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση και γραφειοκρατή γιατί αυτό θα ωφελεί τον κόσμο πιστεύω. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος ε, συνάδελφο το λόγο. Οπότε, παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα τον κύριο Λίντμπεργκ να μας παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω την συντάκτρια, τους ε, εισηγητές. Υπάρχει γενικά συμφωνία ότι είναι σημαντικές οι πόλεις της Ευρώπης όπου μένει το 70% του πληθυσμού και δημιουργείται το 80% του πλούτου. Είναι λοιπόν ε, πολύ ελκυστικά ε, επιχειρηματικά περιβάλλοντα η πώληση και η πόλη επενδύσεων. Οι αστικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αστιφιλίας και της κινητικότητας. Θα πρέπει οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν υψηλή ποιότητα σύστημα μεταφορών που θα καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μεταφοράς ε, ανθρώπων και εμπορευμάτων. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν θέματα όπως συμφόρηση, εκπομπές ρήπων ή χορύπανση. Πιστεύουμε ότι ε, τα οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ισορροπημένο από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Και αυτό είναι το μήνυμα του 2013 για την αστική κινητικότητα ε, και το σχεδιασμό αστικής κινητικότητας. Ε, έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ε, συντονιζόμεθα και συμφωνούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα για ε, ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι 16 ή 17 Ιουνίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών που είναι αρμόδια επί της ουσίας αναμένεται να γίνει στις 13 ή 14 Ιουλίου και αναμένεται ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Έκανα ένα λάθος, με συγχωρείτε. Όχι σκόπιμα όμως, σας βεβαιώνω, να, αφού σας ενημερώσω για τα του φακέλου και τις προθεσμίες, δίνω το λόγο πάλι στην συντάκτρια της νομοδότης, την κυρία Εύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ήταν δύσκολο να περιοριστώ στα όρια που δίνονται για τις γνωμοδοτήσεις. Ελπίζω να ε, έλαβα υπόψη μου όλες τις ιδέες και περιμένω με ενδιαφέρον να συναντήσω και να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνεργασία με τους σκιώδεις. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το, το τελευταίο σημείο για τη, συνα... για τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.